Je vous propose de cesser les conversations particulières et de commencer notre réunion. Σταματήσουμε τις συζητήσεις ε, κατηδίαν και να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίασή μας και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Το σημείο 1 στην ημερήσια διάταξη πρώτα. Όσον αφορά ε, το θέμα των ε, διαρθρωτικών ταμείων είναι ένα ζήτημα το οποίο ήταν αντικείμενο μιας προφορικής ερώτησης, το συζητήσαμε ήδη ε, και στο Στρασβούργο. Υπάρχει και το θέμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τους άστεγους, για τα ζητήματα λοιπόν 17 και 18 σε σχέση με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση θα τα συζητήσουμε σήμερα στις 5 η ώρα γιατί η, Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, ανέβαλε την ε, αυριανή της συνεδρίαση και πρέπει να ε, το λάβουμε αυτό υπόψη πριν από το τέλος σημερινής συνεδρίασης. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη τον, ε, από όσου ε, θα πάρουν ε, το λόγο. Ας πούμε αύριο το πρωί η κυρία Φιγκερέντου θα πρέπει να μην είναι παρούσα γιατί πρέπει να είναι πρόεδρος σε κάποια άλλη επιτροπή. Να ζητήσω συγγνώμη για αυτή την αλλαγή λοιπόν που αναστατώνει κάπως τα πράγματα. Για το σημείο 2 πάντα μεταδίδεται και στο web streaming η συνεδρίασή μας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή για το θέμα της ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας για να μας πει ορισμένα πράγματα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Υπήρξε μια συνεδρία σε ένας τριμερής διάλογος στις 23 Μαΐου και στις την επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είχε μια συνάντηση τη εισηγήτριας που είναι η επικεφαλή για αυτό το χαρτοφυλάκιο με του σκιώδεις εισηγητές τη ΛΥΜΠΕ. Την επόμενη στις 22 Ιουνίου θα υπάρξει ένα τριμερή διάλογος που θα μπορεί να είναι ο τελικός τριμερής διάλογος για να γνωρίζουμε τελικά πώ θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Εγώ αναμένω στι 22 σε αυτό το τριμερή διάλογο να προσκληθεί και να είναι παρούσα η πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης. Ε, γιατί είχαμε μια μακρά μάχη πέρα από θέματα ουσίας για τα δικαιώματα των μεταναστών. Έχουμε μακρά μάχη για να συνεμπλακούμε, όπως λέει και προβλέπει ο κανονισμός, σε ισότιμη βάση με, με την άλλη Κοινοβουλευτική Επιτροπή σε αυτά τα θέματα που εμείς είμαστε η επί της αρμόδια Επιτροπή και αποκλειστικής αρμοδιότητας κιόλας Επιτροπή. Γι' αυτό είχα μια στάση ανοιχτή διαλόγου και αφούγκρασης, ε, αλλά δεν είμαι καθόλου υπέρ του να αντικατασταθεί η θέση της ε, Προέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης ή της εισηγήτριας σε ένα τριμερή διάλογο που πρέπει να εμπλακούμε, μια και είμαστε ουσιοδός αρμόδιοι για τα θεμελιώδη άρθρα αυτής, αυτού του θέματος. Όλα αυτά ήταν πολύ επίμαχα, αλλά πιστεύω οι τελευταίες ειδήσει είναι καλές πρόεδρε και υπάρχει βούληση συνεργασίας πιο ανοιχτή και όχι μόνο για θέματα διαδικασίας αλλά και για θέματα ουσίας επιπλέον. Το θέμα ουσίας που απομένει Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, τα θέματα είναι τρία θέματα που ενέκρινε η ολομέλεια του σώματος μετά από αίτημα της δικής μας επιτροπής. Χάσαμε πολλά αιτήματα, αλλά κερδίσαμε τρία. Και αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο σε αυτά τα τρία θέματα δεν, δεν μας εισακούει. Είναι ένα θέμα ίσονος σημασία ε, που υπάρχει και γλωσσικό θέμα εδώ, αλλά δεν θα υπάρξει ε, πρόβλημα στις αλλαγές ε, για την απασχόληση χρησιμοποιώντας άλλη ορολογία. Όμως το πιο σημαντικό είναι το δικαίωμα των εργαζομένων τρίτων χωρών που εργάστηκαν ή εργαζόντουσαν στην Ευρώπη και επιστρέφουν στη χώρα τους. Και το Συμβούλιο σε περίπτωση που επιστρέψουν στη χώρα τους δεν θα έχουν συντάξεις. Θέλουν να περιοριστεί το δικαίωμα στις συντάξεις. Πρόκειται όμως για ίση μεταχείριση. Πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως και οι κοινοτικοί υπήκοοι. Αυτό είναι ένα θέμα όπου υπάρχει μια κόκκινη διαχωριστική γραμμή. Κόκκινη ιστορική διαχωριστική γραμμή. Και στο Συμβούλιο μόνο ένα κράτος μέλος υποστηρίζει αυτή τη θέση και νομίζω ότι η Επιτροπή ΛΥΒΕ, η Εκτελεστική Επιτροπή, δεν θα πρέπει να υπαναχωρήσουμε ώστε η ίση μεταχείριση να είναι θεμελιώδης αρχή που θα ισχύει για την εξαγωγή και καταβολή των συντάξεων. Ένα άλλο θέμα ίσονος σημασία και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσουμε είναι ότι θέλει το Συμβούλιο η επαγγελματική κατάρτιση για τους ανέργους να περιορίζεται σε εκείνους που έχουν σύμβαση εργασίας πάνω από έξι μήνες. Είναι ένα ίσονος σημασία θέμα αλλά συμβολικό θέμα που έχει και τη σημασία του. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε τέτοιου όρου. Γι' αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε στις του ε, Έχουν οι σάντος, οι σκιώδεις, οι ήδη ενημερωθεί. Δεν υπάρχει κάποια εντολή να ληφθεί κάποια άλλη απόφαση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι θέσει. Εγώ προαναγγέλω ότι αυτή ήταν ε, η ιστορία της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα και μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα ανάλογα με τις επιλογές σας. Ε, θα το δεχτώ αυτό. Αλλά αντίθετα, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θέλει, αν θέλει να απολεστεί κάποιο αίτημα της Επιτροπής Απασχόλησης θα πρέπει πραγματικά να δώσουμε εμείς μάχη για να επιμείνουμε σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά θα ήθελα να σας πω ότι θα σας συνοδεύσω στον επόμενο τριμερή διάλογο και θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Επιτροπής γιατί βάσει του κώδικα ε, που έχουμε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο οι ομάδες, οι διαπραγματευτικές ε, στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων ε, πρέπει να αποτελούνται από τις αρμόδιες επιτροπές. Οπότε επειδή εδώ μιλάμε για συνδεδεμένη ε, επιτροπή. Ελπίζω να μπορέσει να καταλάβει ε, ο Πρόεδρος το αίτημά μας. Μας ζητήθηκε επίσης να εγκρίνουμε την ε, θέση της δικής μας Επιτροπής εν ώψη του επόμενου τριμερούς διαλόγου και βεβαίως μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την απόφαση που λάβαμε για την έκθεσή σας και ε, θα το επιβεβαιώσουμε και μετά το πέρας του τριμερούς διαλόγου και των συμπερασμάτων. Ε, μας, ζητεί, μας ζητάει η Επιτροπή να την υποστηρίξουμε ως το τέλος. Έχετε λάβει επίσης ένα σημείωμα στο φακελό σας για την ακρόαση που είχαμε στις 14 Απριλίου του 2011 με τους κοινωνικούς εταίρους σε σχέση με την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, για την οδηγία για το χρόνο εργασίας και το τελευταίο σημείο ανακοινώσεων του Προέδρου, που είναι επίση σημαντικό, θα θυμάστε, σα είχα επιστήσει την προσοχή στο γεγονό ότι στην Επιτροπή ε, Περιφερειακών Ζητημάτων, στο πλαίσιο τη έκθεση του κυρίου Πίπερ, ε, που είναι η πέμπτη έκθεση συνοχή, για την οποία γνωμοδοτήσαμε και εμείς, η παράγραφος 50 της ε, συγκεκριμένης, 55 διορθώνει ο Πρόεδρος, της ε, συγκεκριμένης έκθεσης, ε, αφορά τις αρμοδιότητες της δικές μας, μπαίνει στα χωράφια τα δικά μας, γιατί ακριβώς αφορά τις συνέπειες παγκοσμιοποίησης. Είχα ενημερώσει εγώ για το θέμα αυτό, γιατί πρόκειται για τη νέα ερμηνεία ε, της, Επιτροπής του, της Επιτροπής ΑΦΚΟ για το άρθρο 50. Η ερμηνεία αυτή εμάς δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνους γιατί ουσιαστικά ε, ε, μια συνδεδεμένη επιτροπή θεωρείται ίση όταν ε, ε, όταν αυτό το επιτρέψει η καθήλυν αρμόδια επιτροπή. Οπότε κατόπιν της έκθεσης της ε, κυρίας Ματιό. Ε, ζήτησα και από τον πρόεδρο Λένε και από τον πρόεδρο ε, Κασίνη μια, μια διευκρίνηση της ε, ερμηνείας του άρθρου αυτού. Όμως το θέμα αυτό δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Βασιζόμαστε λοιπόν στην τρέχουσα ερμηνεία η οποία ουσιαστικά δεν ενεργοποιεί το άρθρο 55 της έκθεσης του κυρίου Πίπερ. Οπότε πρέπει να πούμε ε, να, να ζητήσουμε την υποστήριξη του κυρίου ε, Λένε για να υποστηρίξει τη δική μας ερμηνεία του κανονισμού που επιτρέπει να ε, ισχύουν και οι δικές μας αρμοδιότητες μια συνδεδεμένης επιτροπής που δεν μπορούν καθόλου να παραγνωριστούν. Επίσης, κατόπιν ετήματος της Επιτροπής μας, θα έχουμε μια ξεχωριστή ψηφοφορία για αυτή την παράγραφο 55 και θα ήθελα να καλέσω το σύνολο των ομάδων να κινητοποιηθούν, ώστε οι ομάδες τους, και μιλάω και για το ΕΛΚ, να καταψηφίσουν αυτήν την παράγραφο 55. Τελείωσα με τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μόρτεν Κέρουμ που ε, είναι εδώ σήμερα μαζί μας ε, και υπέστηκε και τις ανακοινώσεις ε, που πρέπει να κάνω στην αρχή της συνεδρίασής μας. Ε, τον καλωσορίζω ως Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει βέβαια αρμοδιότητα που εξεπερνά τις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής, όμως η Επιτροπή μας παρόλα αυτά θέλησε να ακούσει αυτά που ε, έχετε να μας πείτε σε σχέση με την ε, κοινωνική πολιτική, την ε, πολιτική για το χρόνο εργασίας. Είναι κάτι το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων σας και θα θέλαμε να σας ακούσουμε. Επίσης θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε ειδικότερα όσον αφορά την πτυχή των Ρωμά που κινητοποίησε ιδιαίτερα τους πολίτες αλλά και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μάλιστα και ένα ζήτημα αρκετά επί Σα και για σας. Σας δίνω το λόγο κύριε Διευθυντά και μετά ε, θα ακούσετε ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μένα που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και απευθύνομαι σε αυτή την τόσο αξιόλογη ομίγυρη. Ελπίζω ότι αυτή είναι η αρχή μιας πιο συνεχούς επαφής και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στον οργανισμό και την Επιτροπή σας. Όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, έχουμε πάρα πολλά κοινά Σήμερα το πρωί ε, μίλησα στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών ε, και έχουμε αντίγραφα κάποιων ε, εργασιών μας, των δραστηριοτήτων μας και αν θέλετε και άλλα αντίγραφα μπορώ να σας στείλω. Να σας μιλήσω λίγο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις επιτροπές, είναι ένα εγκάσιο θέμα θα έλεγα. Και αυτό για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω εν συντομία όσον αφορά την τρέχουσα εργασία μας είναι τρία θέματα. Το ένα είναι το θέμα των Ρωμά, τα άτομα με, προβλη... με ανάγκες και του, οι μετανάστες ε, που χρησιμοποιούνται για τις οικιακές εργασίες. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα τα οποία άπτονται ε, και της ε, ημερήσιας διάταξης των, την, της δικής σας επιτροπής. Τα μετανάστες, άτομα που επίσης εγκαταλείπουν το σχολείο Ξέρετε, ε, κυρίως όσον αφορά το θέμα των Ρωμά, ότι είναι μια ομάδα ε, η οποία υφίσταται πολλές διακριτικές μεταχειρήσεις. Το 2008 ο οργανισμός μας έκανε μια πανευρωπαϊκή έρευνα, ε, ρώτησε 25.000 άτομα από εθνικές μειονότητες, μεταξύ αυτών και 3.500 Ρωμά και έχουμε επομένως από όλες τις απαντήσεις που πήραμε ένα ε, σημαντικό σημείο που είναι η διακριτική μεταχείριση βάρος των Ρωμά. Σήμερα, σήμερα θα μιλήσω την, για το θέμα της ε, πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου. Ε, όπως ξέρετε, το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα ε, και στο χάρτη αναφέρεται και στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και επομένως το δικαίωμα αυτό ε, πρέπει να το απολαμβάνουν όλοι. Από τις 27 χώρες που έκανε την έρευνα, το, η έρευνα το 2008, η οργανισμός μας, είδαμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ρωμά εγκαταλείπει το σχολείο μετά από πέντε χρόνια ε, σχολικής ζωής. Από, τις, ε, από ένα, αριθμό χωρών ε, είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που εγκατέλειψαν 35-75% των παιδιών εγκατέλειψαν το σχολείο πριν από τα 5 χρόνια και από τον συνολικό αριθμό των παιδιών, είναι λιγότερο από 2% του συνολικού αριθμού των παιδιών που, εγκατέλειψαν τα, που, εγκατέλειψαν το σχολείο, που πηγαίνουν μάλλον στο σχολείο. Επομένω, βλέπουμε ότι επειδή και σε πολλέ σε πολλές περιπτώσει ξεπερνάει και το 75% των, ε, των παιδιών Ρωμά που εγκαταλείπουν το σχολείο, βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ε, ανάμεσα στα, Ρωμά και στα υπόλοιπα παιδιά στο σχολείο και γίνεται η διακριτική μεταχείριση εμφανίζεται με διαφόρους τρόπους. Παραδείγματο χάρη η δημιουργία ειδικών σχολείων για τους Ρωμά, όπου κάπως γετοποιούνται τα παιδιά. Πολλέ χώρε έχουν, έχουν κάνει πρόοδο και έχουν εντάξει ε, τα παιδιά των Ρωμά στην, στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Όμως, εάν δεν γίνουν κάποια βήματα έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε την, την ανεκτικότητα και, την, και, την, το συγχρονισμό, αν θέλετε, όλων των παιδιών στα σχολεία, θα, θα πρέπει να περιορίσουμε επίσης και την εχθρότητα από την πλευρά των εκπαιδευτών ε, και των, ε, του προσωπικού των σχολείων. Ε, δεν θα προχωρήσουμε και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλές φορές τα παιδιά αυτά έχουν να αντιμετωπίσουν και την εχθρότητα των γονέων των άλλων παιδιών. Άρα θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα εδώ. Τώρα, Κάποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να μην συνδέονται άμεσα με θέματα διακριτική μεταχείρισης, αλλά να συνδέονται περισσότερο με κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που επηρεάζουν το σύνολο του πληθυσμού, αλλά και πιο συγκεκριμένα τους Ρωμά. Παραδείγματο χάρη να αναφέρω κάποιους παράγοντες. Δεν είναι ασυνήθιστο η Ρωμά να ε, μένουν σε σπίτια τα οποία δεν συνδέονται, αν θέλετε, με, τις με, την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, παραδείγματο χάρη με τα σχολεία. Επίσης, δεν, μπορεί να, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς. Μπορεί είτε να μην υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς στα σχολεία ή να, μην είναι, ε, να είναι πολύ ακριβή η μεταφορά αυτή. Υπήρχε ένας καταβλισμός Ρωμά, μερικά χιλιόμετρα από το χωριό και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα τα παιδιά αυτά να πάνε στο σχολείο. Δεν υπήρχε λεωφορείο, σχολικό λεωφορείο. Και όταν το, ε, το θίξαμε αυτό το θέμα στον Δήμαρχο, δεν το ήξερε καν, το αγνοούσε το πρόβλημα και ε, μας είπε ότι θα το έβλεπε, διότι οι γονείς των παιδιών μας είπαν ότι η, η, αδυναμία αυτή μεταφοράς, αν θέλετε, ήταν ένα φοβερό μειονέκτημα, ιδίως το χειμώνα. Επίσης, ε, υπάρχει και η πίεση που ασκείται στα παιδιά να μπουν στην αγορά εργασίας πάρα πολύ νωρίς, έτσι ώστε να υποστηρίξουν το οικογενειακό εισόδημα δηλαδή να εγκαταλείψουν το σχολείο και να αρχίσουν να δουλεύουν. Επίσης υπάρχουν και άλλα εμπόδια, πολιτιστικά παραδείγματο χάρη. Οι γονείς μπορεί να μην βλέπουν την συνεισφορά της εκπαίδευσης της παιδείας ε, στον τρόπο της ζωής τους. Επομένως χρειάζεται να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια έτσι ώστε να δούμε αυτοί οι παράγοντες ε, πώς επηρεάζουν την κατάσταση, ποιοι, ποιοι είναι οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες ε, που οδηγούν στη διακριτική μεταχείριση. Γι' αυτό και ο οργανισμός μας κάνει, να κάνει τις μελέτες για την διακριτική μεταχείριση εναντίον των Ρωμά και δεν μελετά μόνο τους Ρωμά, κάνει και έρευνες και με τον πληθυσμό που ζει σε γειτονικέ περιοχές, έτσι ώστε να δούμε πώς ασκούνται τα δικαιώματα ή πώς προφυλάσσονται τα δικαιώματα των Ρωμά. Δηλαδή βλέπουμε τα, κατά πόσον υπάρχει φτώχεια, ε, κατά πόσον υπάρχει διακριτική μεταχείριση για να δούμε και ποιες είναι οι προκλήσεις που ε, υπάρχουν. Ε, έχουμε κάνει ε, επίσης τις έρευνες αυτές με την Παγκόσμια Τράπεζα, με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και βλέπουμε και τι γίνεται και στις άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτά για τους Ρωμά. Τώρα περνάμε στο δεύτερο θέμα που αφορά τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσυπογράψει την ε, Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με ειδικέ Ανάγκες και έχει αναλάβει τη δέσμευση να ε, εξασφαλίσει, να διασφαλίζει τα δικαιώματά τους ελπίζουμε με την έρευνα που κάνουμε και τις μελέτες που κάνουμε ε, να βρούμε τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να ε, προωθήσουμε την θετική διακριτική μεταχείριση και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Εμείς είχαμε ζητήσει και μία πολιτική δέσμευση, διότι είδαμε ότι κάποια κράτη-μέλη εφαρμόζουν μια γενική εξαίρεση ε, για τα άτομα τα οποία έχουν πνευματικές αναπηρίες ε, ή έχουν κάποια άλλα προβλήματα όσον αφορά τις, τα εκλογικά τους δικαιώματα. Και ε, σε 7 κράτη-μέλη κάτι τέτοιο ισχύει. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν μελετήσει την έκθεσή μας και προσπαθούν να προσαρμόσουν την νομοθεσία τους στο σημείο αυτό, διότι πραγματικά ε, δεν μπορεί να δεχτούμε τον αποκλεισμό ε, των ατόμων αυτών από την πολιτική ζωή και από την δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέσσερα θέματα μας απασχολούν εδώ. Το ένα είναι οι συνθήκες ε, σε μακροπρόθεσμα σε κάποια ιδρύματα, σε διάφορους οίκους ε, ευγυρίες ή οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον είναι η νομική τους ικανότητα. Τρίτον είναι η συμμετοχή τους στις κοινωνικές δραστηριότητες. Και ε, τέταρτον η πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη ο οργανισμός μας θα δημοσιεύσει μία μελέτη που στηρίζεται σε διάφορες συνεντεύξεις που πήραμε σε εννέα χώρες και που βλέπουν ποια είναι η κατάσταση επιτόπου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συλλέξουμε συγκρίσιμα στοιχεία για πολλά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ιδρύματα σε όλες τις 27 χώρες και ακριβώς επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε ιδρύματα. Ίσως είναι και λιγότερο σημαντικό να μην εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάποια ιδρύματα πράγματα, αυτά καθεαυτά, αλλά περισσότερο να αλλάξουμε την φιλοσοφία πώς δηλαδή οι φροντίδες προσφέρονται σε αυτά τα ιδρύματα. Να μην υπάρχει μία μεταχείριση γενική, ε, αλλά να ε, προσπαθούμε να τα εντάξουμε τα άτομα αυτά στην κοινωνία. Να σας πω ποια είναι τα τέσσερα θέματα τα οποία ε, προκύπτουν από, την αρχική μας μελέτη, αν θέλετε. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Καταρχάς, η αποϊδρυματοποίηση ε, είναι ε, κάτι το οποίο προωθούμε. Θέλουμε να υπάρξει μια να, να, να είναι ανεξάρτητα τα άτομα αυτά και να ζουν στην, ε, στην κοινωνία. Βέβαια, θα πρέπει οι διαδικασίες αυτές να είναι πολύ καλά συντονισμένες. Δεν είναι απλώς και μόνο ε, δεν αρκεί απλώς και μόνο να κλείσουμε ένα ίδρυμα και από εκεί και πέρα να βγάλουμε τα άτομα αυτά στο δρόμο από τη μια μέρα στην άλλη. Είδαμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη έγινε αυτό και τι έγινε. Ε, είδαμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να ε, πετύχουμε. Άρα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια πολύ ε, ευαίσθητη ισορροπία εδώ, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε. Δεύτερον, οι ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει να ε, χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να αναπτύξουμε την, τις δυνατότητες να ζουν ανεξάρτητα άτομα αυτά και όχι να ζουν μέσα σε ιδρύματα. Τρίτον, οι μελέτες μας απέδειξαν ότι τα άτομα με αναπηρία ε, θεωρούν ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν κάποια απασχόληση, κάποια δουλειά. Ε, σε προσωπικό επίπεδο αυτό τους προσφέρει ένα νόημα στη ζωή τους. Ταυτόχρονα, και αυτό μας εκπλήσει βέβαια, και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να τα προφυλάξουμε τα άτομα αυτά από τον κίνδυνο εκμετάλλευση ε, από κάποιους άλλους που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ε, σαν δωρεάν ε, εργατικά χέρια. Κάποιο μας είπε ότι το σπίτι του διευθυντή ενό ιδρύματος χτίστηκε χρησιμοποιώντα την δωρεάν εργασία των ατόμων που φιλοξενούσε το ίδρυμα. Επίσης, ε, το οργανισμός μας ε, είδε ότι ε, ο καλύτερος τρόπος για να ανοίξουμε την αγορά εργασίας στα άτομα αυτά είναι να τους επιτρέψουμε να μπουν στο εκπαιδευτικό σύστημα προσφέροντάς τους μια all-inclusive, αν θέλετε, εκπαίδευση. Επομένως, πιστεύουμε ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ε, γυρίζουν σελίδα. Ε, αλλάζουμε τελείως ε, την οπτική αντιμετώπιση τους, εστιάζουμε την προσοχή μας στο άτομο και όχι στην αναπηρία. Και πιστεύω ότι τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα πάρα πολύ ενδιαφέροντα για μας. Τώρα, να μιλήσω ε, και για την εργασία του οργανισμού μας ε, στα θέματα των μεταναστών και της, οικονομική, και της χρησιμοποίησής τους για τις οικιακές εργασίες. Υπάρχει μία μελέτη η οποία αφορά τους νόμιμους μετανάστες και αφορά τους υπαλλήλους, τους συγγνώμη, μετανάστες τρίτων χωρών που ε, απασχολούνται σε οικιακές εργασίες δεν ασχολούμεθα με άτομα τα οποία εργάζονται παραβιάζοντας τις διατάξεις για τη βίζα. Κάναμε μία έρευνα σε 10 κράτη-μέλη, κάναμε συνεντεύξεις με διάφορους εργαζόμενους και με διάφορες οργανώσεις ε, της ε, πολιτών και ε, έγινε μια πρώτη προσπάθεια να αναλύσουμε την ε, κατάσταση που επικρατεί σε μερικά κράτη-μέλη και εξετάσαμε τους, τους ε, συνθήκες εργασίας, την, την ελευθερία του να δημιουργούν οργανώσεις, την οικογενειακή τους ζωή και θα αναφερθώ σε τρεις προκλήσεις αν θέλετε που ανακαλύψαμε. Καταρχάς μιλάμε για μια ομάδα που είναι πολύ εύκολο να υποστεί διακριτική μεταχείριση. Οι περισσότερες είναι γυναίκες. Επομένως, έχουμε και τα θέματα φιλετικών διακρίσεων, διακρίσεων λόγω του φίλου. Η σεξουαλική παρενόχληση και η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος. Επίσης, ε, οι γυναίκες αυτές είναι ευάλωτες λόγω ακριβώς και της, της φιλετικής τους προέλευσης σε καμιά φορά. Επίσης υπάρχει και ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την σύμβαση ε, του Διεθνού Γραφείου εργασία όσον αφορά τις, ε, ε, εργαζόμενους στα σπίτια, τις οικιακές βοηθούς. Επίσης υπάρχουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων αυτών στην δικαιοσύνη όταν θέλουν να καταγγείλουν την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Ε, ο κίνδυνος, ε, ο φόβος τους μάλλον είναι ότι εάν στραφούν στις αρχές θα τους ε, καταγγείλουν οι εργοδότες τους στην στις, μετανάστευση. στις υπηρεσίες μετανάστευσης. Τώρα, εάν υπάρχουν παράνομοι μετανάστες στην αγορά εργασίας, αυτοί οι άνθρωποι εποφελούνται από τα ίδια δικαιώματα, ε, τα, δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στις ευρωπαϊκές συμβάσεις, στις συμβάσεις του, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας κτλ. Εκτός και αν οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν κάτι διαφορετικό. Ουσιαστικά το, η εθνική νομοθεσία δεν ε, εγγυάται ρητά κάτι τέτοιο και θα αναφερθώ σε δύο γνώμες που έχουμε. Καταρχάς ε, είναι η εισαγωγή ε, ε, συγκεκριμένων διατάξεων όσον αφορά την ελάχιστη αμοιβή, στις, την αποζημίωση για ατυχήματα, την ασφάλεια υγείας κτλ. Και τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ζήτηση για, αυτά τα, για αυτές τις θέσεις, αν θέλετε, για αυτά τα άτομα και θα μπορούσαν ε, μέσω μεταναστευτικής πολιτικής ε, να ε, νομιμοποιήσουν τα άτομα αυτά και να, έχουν, να, να χαίρουν μεγαλύτερης προστασίας οι πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρώμα, τα άτομα με ειδικέ ανάγκε και η οικιακή βοηθή, δείχνουν πόσα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αυτών, ακριβώ όπως αναφέρονται στη Σύμβαση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, η Επιτροπή σας ε, έχει την ε, ικανότητα να βοηθήσει στο έργο μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Είμαι έτοιμος να δεχτώ τις ερωτήσεις σας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά για αυτή την τόσο συγκεκριμένη παρουσίαση των προβλημάτων που απασχολούν τα άτομα αυτά και που μας απασχολούν και εμάς. Ο κύριος Αλέξανδρος Σάρκας πρώτα και μετά η κυρία Ελίζαμπετ Σρότερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Διευθυντά. Και ξεκινάω ευχαριστώντας σας. Όχι μόνο για τα πρακτικά, αλλά επειδή πολύ ειλικρινά με τα τελευταία σας λόγια αποδείξατε ότι αξίζει η υπηρεσία σας και το άτομό σας στο έργο σας όταν αναγνωρίζετε το στρατηγικό έργο, η σημασία αυτού του έργου σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Εγώ πιστεύω και το συμμεριζόμαστε αυτό, ότι η αξιοπρέπεια μιας κοινωνίας δεν μετράται μόνο στο ΑΕΠ το εισόδημα ανακεφαλήν, που στατιστικά βλέπουμε ποιο είναι αλλά από το σεβασμό που έχουμε για τους πιο ευάλωτους, για εκείνους που συμβιώνουν μαζί μας και είναι πιο ευάλωτοι. Και πώς μπορούμε συλλογικά να βοηθήσουμε εκείνοι που δεν έχουν τα μέσα για να πετύχουν μια αξιοπρεπή ζωή, να βοηθηθούν και να μην αγνοηθούν από τους άλλους πολίτες, από την υπόλοιπη κοινωνία. Να απλώσουμε το χέρι μας και να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό έχω κάποιες ερωτήσεις, κύριε Γενική Διευθυντά αξιολογώντας και εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο σας ε, και για τις ε, προοπτικές ε, που έχετε, θα ήθελα να ξέρουμε αν άρχισαν και έγιναν ή αν υπάρχουν κάποιες μελέτες που αποσαφηνίζουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα το ότι δεν μπορούν να διαφοροποιούνται σε σχέση με αν είναι κάποιος πολίτης μιας κοινοτικής χώρας ή πολίτης μιας έξω χώρας. Και εδώ η πολιτης μιας εξωκοινοτικης χωρας και ίδια και τα δικαιώματα είναι τα ίδια για όλους τους πολίτες που ζουν στην Ευρώπη και όχι μόνο για τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό, διότι εγκρίνουμε νομοθετικό έργο, μέτρα κατά της αρνητικής μεταχείρισης και όταν έρχεται η ώρα της αλήθειας βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες πολίτες στην Ευρώπη. Παρότι κάνουμε λόγο για τη μη αρνητική μεταχείριση, εκείνη που είναι εκτός Ευρώπης και δεν κάνω λόγο για τους παράνομους, αλλά για εκείνους που βρίσκονται νόμιμα ανάμεσά μας. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση βάρο βάρος λοιπόν και είναι πολίτε δεύτερη κατηγορία. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση ανάλογα με την άδεια που έχουν άδεια παραμονής ή σύμβαση εργασία ή προέλευση. Και ένα τελευταίο ερώτημα επίση Είναι προφανέ ότι τον 20ο αιώνα <clears throat> προχωρήσαμε όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι δηλαδή επεκτείνονται αυτά τα δικαιώματα και έχουμε και δικαιώματα δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, δικαιώματα κοινωνικά, δικαιώματα οικονομικά. Όχι μόνο το πρώτο, ας το πω έτσι, κεκτημένο των δικαιωμάτων, αλλά και επέκτασή τους. Η υπηρεσία σας είναι σε θέση να επεκτείνει λοιπόν αυτές τις έννοιες, ώστε να υπάρξει μια πολύ ευρύτερη έννοια όσον αφορά την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και για το αν μπορεί και εργάζεται, πώς μπορεί να καταρτιστεί, να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος, το άτομο. Ευχαριστώ. κυρία Σρέτερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα βρήκα την ε, ενημέρωσή σας. Θα κάνω μια επιμέρους παρέμβαση και μια γενικότερη φύσεως. Σε ό,τι αφορά την έκθεση για τα άτομα με αναπηρίες, είναι πολύ ωραίο ότι θα ανοίξουν τα σχολικά συστήματα. Πρώτα θα γίνει αυτό και μετά ενδεχομένως θα διασφαλίσουμε ε, το άνοιγμα και της ε, κύριας αγοράς εργασίας. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν και οι αντίστροφες διαδικασίες βέβαια. Εγώ είμαι υπέρ της δικής σας προσέγγισης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως Έχουμε το πρόβλημα ότι υπάρχει μαζικός αποκλισμός ε, στο Συμβούλιο ενάντια στην πέμπτη οδηγία κατά των διακρίσεων που ασχολείται με αυτό το θέμα και που μέσα από τις τροπολογίες μας ε, θα γίνει η ευρωπαϊκή εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Ξέρουμε ποιος μπλοκάρει και ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο αποκλεισμός του κειμένου. Με ενδιαφέρει όμως εσείς τι κάνετε για να έρθει το εμπάργο αυτό στο Συμβούλιο. Έχω την εντύπωση ότι στη Γερμανία υπάρχουν κάποιες σχετικές κινήσεις ε, γιατί είναι αρμόδια τα ομόσπονδα κρατήδια και όλο και περισσότερα θέλουν να αναπτύξουν ένα σύστημα χωρίς ε, αποκλεισμούς. Ε, τι υποστήριξη παρέχετε εσείς. Υπάρχει και η ΠΕΜ, τη Οδηγία κατά των Διακρίσεων, αλλά και άλλοι ε, δρόμοι για να επιτύχουμε το στόχο μας. Εσείς τι πιστεύετε. Εμείς νομίζουμε ότι η πέμπτη οδηγία κατά των διακρίσεων είναι ο μοναδικός σωστός δρόμος και θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Ένα ήταν αυτό. Το άλλο πολύ σύντομα. Κάποια κράτη-μέλη απαλλάχτηκαν, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, από την πλήρη εφαρμογή στο εσωτερικό δίκαιο της ε, ε, οδηγίας ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υποστήριξη θυμάτων και ομαδική προσφυγή. Εσείς ε, εξετάσατε τι συνέπειες θα προκύψουν στα κράτη-μέλη όπου δεν προβλέπετε σύστημα συλλογικής προσφυγής. Κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών. Ε, βλέπω ότι όλοι, ναι, όλοι έχουν ζητήσει, ε, βρίσκονται εδώ όσοι βρίσκονται εδώ έχουν ζητήσει το λόγο. Τώρα η κυρία Λίνε. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζοντας αυτό που είπε για την οδηγία, για, την ανα, τις αναπηρίες ε, που έχει κολλήσει το Συμβούλιο, όπως είπε η κυρία Σρόντερ, θα θέλαμε... Ξέρουμε δηλαδή ποια είναι τα κράτη-μέλη που δημιουργούν το πρόβλημα. όσον αφορά το θέμα της έκθεσης που είπατε ότι θα ε, δημοσιευθεί την ε, επόμενη χρονιά. Εγώ θα ήθελα να μάθω ε, τα διαρθρωτικά κονδύλια στις χώρες τις οποίες εξετάσατε πώς όντως αξιοποιήθηκαν στον τομέα της φροντίδας στο πλαίσιο, μιας, στο πλαίσιο της κοινωνίας. Και κάτι ακόμη, Μιλήσατε επίσης ε, για τα προβλήματα διανοητικής καθυστέρησης και τα προβλήματα ανθρώπων με δυσκολίες εκμάθησης. Ε, στα Ινστιτούτα ε, τι είδου εξοπλισμός υπάρχει Και μερικές φορές μάλιστα ε, χρησιμοποιούνται αυτά τα cage beds ε, που ε, ουσιαστικά σκοπό έχουν να περιορίσουν κάπως τα, τα άτομα αυτά. Πριν από πολλά χρόνια είχαμε μιλήσει για τα ζητήματα κινητικότητας και ευχαίρομαι που ε, ορισμένα πράγματα έχουν προχωρήσει από τότε. Υπάρχει όμως και το θέμα των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Υπάρχει μία έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί, αλλά θα εξετάσει τα ζητήματα ε, των ε, ηλικιωμένων. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να δούμε κατά πόσο η κοινωνία αρνείται τα θεμελιώδη δικαιώματα μιας ε, ομάδας ανθρώπων όπως είναι οι ηλικιωμένοι. Έγινε και μία διάσκεψη σήμερα για τους ηλικιωμένου ανθρώπους που δεν ε, συμμετέχουν σε ε, κλινικές δοκιμές παρά το γεγονός ότι τα φάρμακα που θα προκύψουν από τις δοκιμές αυτές θα χρησιμοποιηθούν για ηλικιωμένου ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα άρνησης θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπάρχουν και άλλες πτυχές που πρέπει ακόμη να εξεταστούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόντο και μετά θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε κύριε Κέραμ. Η κυρία Κόζα. Ο, ο κύριος Κόζα, συγγνώμη. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση αλλά επειδή ένα τμήμα όσων ήθελα να πω υπόθηκε ήδη, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την δουλειά του οργανισμού σας ως σήμερα και θα ήθελα να σας πω επίσης ότι είμαι ο εισηγητής της έκθεσης για τα άτομα με αναπηρίες. Καταλαβαίνετε ότι γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες. Ε, ο οργανισμός σας έχει σκοπό να ε, εκπονήσει μια σφαιρική μελέτη για τα ζητήματα αυτά. Και θα ήθελα επίσης να μάθω σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται η συνθήκη της Λισαβόνας ε, και τώρα Αναφέρομαι κυρίως στο βαθμό στον οποίο ε, συμμορφώνεται με την σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα, το δικαίωμα ε, ψήφου των ανθρώπων με ε, πνευματική αναπηρία, η συμμετοχή τους στο πολιτικό βίο. Είναι ένα ζήτημα που επίσης θα ήθελα να θέσω. Και θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν θα διευρύνεται το πεδίο εξέτασης ώστε να μην συμπεριλαμβάνει έννοια άτομα με αναπηρίες μόνο τα άτομα ε, με πνευματική αναπηρία. Υπάρχουν και άτομα με άλλου είδους αναπηρίες. Όσον αφορά τώρα τη χρήση της μητρικής γλώσσας, προβλέπετε να γίνει κάποια έρευνα σε σχέση με τους ε, ανθρώπους που μιλούν στη νοηματική γλώσσα. Πώς μπορούν λοιπόν να έχουν δικαιώματα ε, επικοινωνίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να απαντήσετε στις τέσσερις αυτές ερωτήσεις ε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται, γιατί θα έχουμε και άλλες ερωτήσεις μετά. Um, Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν για το ζήτημα των διαφορών εις ό,τι αφορά την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα βασικά δικαιώματα τα έχουν όλοι, τα απολαμβάνουν όλοι και τα δικαιώματα του χάρτη και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και ε, όλοι ε, προβλέπουν τα ίδια δικαιώματα, είτε πρόκειται για όλες τις κατηγορίες των ε, αλλοδαπών. Και μετά υπάρχουν και δικαιώματα που δεν τα απολαμβάνουν οι μη υπήκοοι. Μετά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κινούμαθα εκτός από το καθεστώς που διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από... Και καλύπτει τουρίστες, προσωρινώς εργαζομένους, ε, μόνιμα διαμένοντες και διαφορά και μετά οι η Η διαφοροποίηση συνήθως είναι μέσα στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από την πλευρά των διακρίσεων αυτό είναι κάτι που το λαμβάνουμε συχνά υπόψη και το αναφέρουμε στις εκθέσεις μας. Αλλά εκεί μπορούμε να το συζητήσουμε και σε διμερές επίπεδο. Ε, δηλαδή αν θέλετε να μπω σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες που έχετε υπόψη σας. Τώρα, για το γενικότερο ζήτημα της οριζόντιας οδηγίας και τα, το, το, το μπλοκάρισμα που γίνεται στο σύστημα. Ε, ο οργανισμός δεν έχει εντολή να παρεμβαίνει άμεσα στην πολιτική και διαδικασία, αλλά καταρτίζουμε πολλές εκθέσεις για τις αναπηρίες, για το σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλα δικαιώματα που έχουν σημασία για την οριζόντια οδηγία. Ξέρω ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ και στα επιχειρήματα και στις συζητήσεις, τα στοιχεία τα δικά μας δηλαδή. Ε, και αυτή είναι η καλύτερη συμβολή του οργανισμού για να καταδείξουμε το πρόβλημα και να ε, εντοπίσουμε την ύπαρξη ενός νομικού κενού που καλό θα ήταν να αντιμετωπιστεί και να κλείσει. Και βέβαια θα ήμουν πολύ ευτυχής να εργαστώ μαζί με την Επιτροπή σας και σε διμερές επίπεδο αν υπάρχουν επιμέρους μελέτες. που θα δώσουν συμπληρωματικά στοιχεία για να εξεταστούν, για να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμβάλλουμε κι εμεί. Τώρα για τη συλλογική προσφυγή πρέπει να πω ότι αυτό δεν μας απασχόλησε συγκεκριμένα, αλλά έχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη και παράλληλα με αυτό ε, συζητούμε και το θέμα της ε, συλλογικής ή ομαδικής πρόσφυγης. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε αργότερα καλύτερα. Για τα διαρθρωτικά ταμεία και πώς χρησιμοποιούνται αυτά, ε, ε, διαισθάνομαι ότι γνωρίζετε πολύ καλά. Δηλαδή κατάλαβα ότι γνωρίζετε... Ό, όχι, ε, γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα των διορθωτικών ταμείων και το κίνημα των αναπήρων το εντοπίζει είχαμε κάποιες άτυπες συνομιλίες με ορισμένους αξιωματούχους και εκεί σημειώνονται εξελίξεις. Αλλά υπάρχουν και περιορισμοί βέβαια σχετικά με τη χρήση ή μη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Πάντως υπάρχει επίγνωση των ταμείων και της λειτουργίας τους και είναι πάρα πολύ χρήσιμη και η σύμβαση για να ε, δούμε αυτές τις ε, συνιστώσεις του προβλήματος. Τώρα για αυτά τα κρεβάτια κελιά, αν θέλετε, που περιορίζουν πολύ τους τροφίμους, ε, δεν το ξέρω το θέμα, αλλά το επεξεργαζόμαστε μαζί με συναδέλφους οι οποίοι συντάσσουν η έκθεση. Ε, γι' αυτά λοιπόν τα κρεβάτια κελιά ή κλουβιά... Ε, θα εκπλησόμουν πολύ αν δεν μας απασχολούσε αυτό το θέμα. Ε, τώρα συνεργαζόμεθα στενά για την σύνταξη της έκθεσης με ανθρώπους με αναπηρίες και ψυχικά προβλήματα για να είμαστε βέβαιοι ότι θα πιάσουμε όλα τα σημαντικά για εκείνους προβλήματα σε επίπεδο κρατών μελών. Και αυτό πραγματικά μας άνοιξε τα μάτια σε πολλούς από εμά σχετικά με την κατάσταση και το μέγεθος των προκλήσεων. Ε, δεν ε, Μιλήσαμε ειδικότερα, δεν καταπιαστήκαμε ιδιαίτερα με την κατηγορία των ηλικιωμένων, αλλά δεν αποκλείω να κάνουμε κάτι περισσότερο εδώ στο μέλλον. Πάντως θεωρούμε ότι όταν ασχολούμεθα με το, τον τρόπο λειτουργίας των ε, ιδρυμάτων, όταν μετακινούνται τα ιδρύματα σε μια πιο εξατομικευμένη και όχι ιδρυματική γενικότερη προσέγγιση, τότε μπαίνει στο επίκεντρο το συγκεκριμένο πρόσωπο και όχι τη ιδρυματική πολιτική. Βέβαια δεν είναι τα πράγματα άσπρο-μαύρο, αλλά θα υπάρξει αλλαγή και εδώ και θα υπάρχουν και παρεπόμενα ωφέλη, αν θέλετε, σε άλλα ιδρύματα. Θα αρχίσουμε ας πούμε, να δουλεύουμε στρατηγικά σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι θα έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο. Ε, γιατί αυτός είναι ο τρόπος αντιμετώπισης ε, των ανθρώπων που είναι στα Ιδρύματα, είτε πρόκειται για μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, ανάπηρους κλπ. Αλλά οπωσδήποτε οι ηλικιωμένοι είναι ένα θέμα το οποίο μπαίνει στην ημερήσια διάταξή μας. Τώρα για το δικαίωμα παθητικής ε, συμμετοχής σε εκλογές, το δικαίωμα του εκλέγην όταν υποβάλαμε την έκθεση και μετρήσαμε τις αντιδράσεις, είδαμε θετικές αντιδράσεις σε αρκετά γιατί αρκετοί είπαν δηλαδή ότι «Α, εδώ είναι, υπάρχει ένα θέμα που δεν το είχαμε σκεφτεί». Χρειάζεται η νομοθεσία όμως που δεν υπάρχει, γιατί δεν είχε προβλεφθεί. Κανείς δεν είχε ε, επικεντρωθεί στο ζήτημα αυτό. Ενώ τώρα με την έκθεσή μας υπάρχει αυξημένη εστίαση στο πρόβλημα και αυτό ελπίζω ότι θα επηρεάσει και άλλες ομάδες που επίσης ε, αποκλείονται τώρα από την πολιτική συμμετοχή και οπωσδήποτε θα το παρακολουθήσουμε το θέμα για να δούμε αν ε, γίνονται αυτόματα τα πράγματα ή αν χρειάζονται καινούριε εκθέσεις. Αλλά οπωσδήποτε και αυτό θέλω να το συζητήσουμε μαζί εμείς για να έχουμε μια αίσθηση της τάξης μεγέθους του προβλήματος. Τώρα για τη μητρική γλώσσα, τη νοηματική γλώσσα, εδώ και αυτό είναι ένα θέμα που θα συμπεριληφθεί στις εργασίες μας. Δεν ε, το έχουμε τώρα, αλλά ε, θα το αντιμετωπίσουμε στις μελλοντικές μας εργασίες. Δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα ενεργού συμμετοχής επίσης, όχι μόνο σε πολιτικές διαργασίες, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους τέσσερις τελευταίους ομιλητές, ζητώντα τους να είναι όσο το δυνατόν ε, λογικότεροι, όπως και η πρώτη. Πρώτα η κυρία Μπλικεβιτσίτα και μετά η κυρία Σεσλοβένσκα. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Διευθύντα για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε για το έργο σας στον τομέα των συγκάνων και των ατόμων με αναπηρίες τους εργαζομένους ε, από τρίτες χώρες. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχετε κάποια στοιχεία στην επισκόπησή σας, στη διάθεσή σας για το πώς τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία έχουν κάποια επίπτωση σε άτομα με αναπηρίες. Είχαν επίπτωση στην ε, ένταξή τους, στην κοινωνική των ατόμων με αναπηρίες, γιατί έχουμε περιπτώσεις στα κράτη-μέλη όπου υπήρξαν περικοπές κονδυλίων δημοσιονομικά σε σχέση με την ένταξη ατόμων με αναπηρίες. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά ε, την, ε, το θέμα των μεταναστών εργαζομένων. Στην ανάλυση σας εντοπίσατε, είδατε ποια είναι η προσέγγιση και η αντιμετώπιση όσον αφορά τα κράτη-μέλη απέναντι σε αυτά τα άτομα, ιδιαίτερα με την αύξηση της ανεργίας που υπάρχει, υπάρχει κάποια αρνητική διακριτική μεταχείριση σε σχέση με εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. E, ήθελα, θα ήθελα να πω ότι οι απαιτούνται λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα έχοντας μια καλύτερη πολιτική η χειρότερη πολιτική δίνονται ανάλογα διαφορετικές απαντήσεις στην κοινωνική πολιτική. Πολλές φορές ε, δεν εξετάζονται ε, θέματα κοινωνικής ε, υποστήριξης, κοινωνικής αρρωγής και ιδιαίτερα δημιουργούνται πρόβλημα για την οικογενική ζωή και τα παιδιά κιόλα. Έχετε κάποιες ενδείξεις όσον αφορά την ευημερία, το επίπεδο ε, των δυνατοτήτων των παιδιών απέναντι στις υποχρεώσεις ε, που έχουν στα παιδιά τους και πώς ανταποκρίνονται μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Και όσον αφορά άτομα που είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, και δεν, υλοποιούν, ε, δεν μπορούν να υλοποιήσουν και να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Κάτι θα έπρεπε να κάνουμε σε σχέση με αυτή την κατάσταση, ώστε οι γονείς και η κοινωνία να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Διευθυντή που μας διαφώτισε για όλα αυτά τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ερώτηση μου είναι σχετική με αυτή που έκανε η συνάδελφος πριν από λίγο. Περιγράψατε λεπτομερώς την κατάσταση που αφορά τα παιδιά των Ρωμά που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και μιλήσατε για την απομόνωση αν θέλετε από τη μια και από το, το, το, ε, το μη σεβασμό του δικαιώματος ε, για εκπαίδευση, Έχετε κάνει ανάλυση ε, της κατάστασης ε, σε κάθε χώρα όσον αφορά τα project που αφορούν την ε, ένταξη των παιδιών αυτών ε, στην σχολική ζωή, στην κοινωνία εν γέννη και στην αγορά της εργασίας. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω το Διευθυντή. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή εδώ. Ε, μια γενικότερη ερώτηση καταρχήν και αν το είπατε αγνοήστε την. Προφανώς ε, εσείς θέλετε να εφαρμόσετε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και ένα πράγμα που μας είπαν μετά τη Λισαβόνα είναι ότι ε, εδώ θα κάνει διαφορά. Ε, πώς δηλαδή, στην πράξη τι διαφορά σημειώθηκε, ενίσχυσε ας πούμε τις αρμοδιότητές σας, ε, τον οργανισμό σας, ποια ήταν η διαφορά. Δεύτερον, για τους οικιακούς εργαζομένους. Ένα από τα θέματα που μας δυσκολεύει εδώ είναι ότι κάποιοι, αν όχι όλοι, εργάζονται σε οικογένειες. Μιλήσατε για σαφή πρότυπα και μία πρόταση που υποβάλαμε εμείς στην εκθεσή μας ήταν να δούμε υποδειγματικές συμβάσεις σε εθνική περιφερειακή βάση. Μπορείτε να μας, να μας πείτε λεπτομέρειες. Δηλαδή, το γεγονός ότι είναι ας πούμε, στο σπίτι μιας οικογένειας αυτό δημιουργεί εντάσεις κλπ. Πώς το βλέπετε το θέμα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, για την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και τον αντίκτυπο που έχει και σε άτομα με αναπηρία και σε υπηκόους τρίτων χωρών. Στις δικές μας τις έρευνες δεν μπορούμε να το δούμε αυτό γιατί ο οργανισμός είναι ακόμα νεαρότατος. Δημιουργηθήκαμε το 2007 και έπρεπε να σιγά σιγά να προχωρήσουμε. Τώρα βλέπουμε τις πρώτες μελέτες σε έναν αριθμό αποτομής και ελπίζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα επαναλάβουμε κάποιες μελέτες μας και τότε θα αρχίσουμε να εντοπίζουμε τάσεις και να πούμε «Α, εδώ διαγράφεται ένα σαφές ε, χαρακτηριστικό της οικονομικής κρίσης ή οτιδήποτε». Ελπίζουμε ότι θα δούμε και άλλα χαρακτηριστικά που θα έχουν επηρεαστεί από αλλαγή στην νομοθεσία, πολιτικές προπρωτοβουλίες που θα αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα. Ιδρυθήκαμε λοιπόν στο δεύτερο Α, δημιουργήσαμε το Radar, μια μικρή μονάδα, στις αρχές του 2008 όταν ε, είδαμε να έρχεται η κρίση για να δούμε τον αντίκτυπό της. Τα άτομα με αναπηρίες ε, δεν είχαν συμπεριληφθεί σε μελέτες, ούτως ώστε να έχουμε κάποια αρχικά στοιχεία και να δούμε τις εξελίξεις μετά. Πάντως, οπωσδήποτε, ε, είναι πιθανότατο ότι θα επηρεάστηκαν από την κρίση δυσμενός. Επίσης φαίνεται ότι ε, ήταν καταλήτης για κάποιες αλλαγές, γιατί ναι μεν πρέπει να εξοικονομούμε χρήμα, αλλά θα πρέπει να εξορθολογικοποιούμε και τα συστήματά μας. Α, τώρα σε ποιο βαθμό θα... Ε, εξελιχθούν αυτά δεν ξέρω γιατί έκανα μόνο κάποιες προσωπικές συζητήσεις. Θα δούμε. Τώρα για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες, ε, εδώ πιο ξεκάθαρα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Πολλοί από αυτούς τους εργαζομένους που δουλεύουν είτε στην κρίζα είτε στη μαύρη οικονομία, ακόμα να είναι σε εκκρεμότητα. Υπάρχουν στοιχεία που πήραμε και δείχνουν ότι οι απολυμμένοι, ας πούμε, στον ε, τομέα των οικοδομών κλπ. Ε, δεν βρίσκονται, δηλαδή δεν ε, καλύπτονται από τον αριθμό των ατόμων που νομίμως αποχώρησαν. Οπότε αυτή είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης ίσως. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια αγορά εργασίας σε ορισμένους τομείς με πολύ υψηλό δίκτυ εκμετάλλευσης. Ε, αυτών των ανθρώπων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το ψάξουμε πολύ καλύτερα το θέμα το 2013 στα πλαίσια του προγράμματος εργασιών μας για να ετοιμάσουμε κάποιες μεθοδολογίες αντιμετώπισης του θέματος. Τώρα για τα προγράμματα ε, ενσωμάτωσης και τις υποχρεώσεις των γονέων απέναντι στα παιδιά τους είναι ένα θέμα, όπως είπα, σε σχέση με τους Ρωμά αυτό. Και πρέπει να πούμε ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αυτό είναι βασικό δικαίωμα όλων των παιδιών, δηλαδή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και μετά θα πρέπει να τα δούμε αναλυτικότερα. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάποια παιδιά δεν πάνε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί συμβαίνει αυτό γιατί είναι, έχουν διακριτική μεταχείριση που αντιμετωπίζουν, γιατί είναι φτωχοί, γιατί φταίνει οι γονείς. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί το μικρό παιδάκι έχει ε, απόλυτο δικαίωμα στην εκπαίδευση και είναι υποχρέωσή μας να δούμε εμείς ως κοινωνία πώς θα παρέμβουμε και θα φροντίσουμε ώστε το κάθε παιδί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Είναι περίπλοκο και καθόλου εύκολο το θέμα αυτό, όμως πρέπει να σηκώσουμε το γάντι. Στην ανακοίνωση της Κομισιόν, ο οργανισμός καλείται να αλληλεπιδράσει με τα κράτη-μέλη σε επίπεδο εθνικών στρατηγικών με βάση τις μελέτες, τις έρευνές μας και τα πορίσματά μας και μετά να ε, αλληλεπιδράσουμε σε επίπεδο εθνικών στρατηγικών και να κάνουμε και πειράματα μεθοδολογικά σε πιλωτικό επίπεδο ούτως ώστε να προσφέρουμε εργαλεία αντιμετώπισης και ορθές πρακτικές. Τώρα, η συνθήκη της Λισαβόνας και αν αυτή επηρέασε θετικά. Η συνθήκη της Λισαβόνας νομίζω ότι έδωσε τεράστια όθηση σε όλον τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά βελτιώνονται πολύ έντονα αυτά τα χρόνια μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Και ο οργανισμός σαφώς εντοπίζει αυξανόμετη επίγνωση, συνειδητοποίηση των ε, υποχρεώσεων στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τους εργαζόμενους στα σπίτια, ε, ε, όταν θα κατατεθεί η έκθεση, θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε, γιατί ανάλογα με τα πορίσματα της έκθεσης ε, θα δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Ε, νιώθω ότι με πιέζει ο χρόνος, πρέπει να τελειώνω και εδώ είναι σύνθετο το θέμα γιατί πράγματι δουλεύουν μέσα σε μια οικογένεια και πόσοι θα θέλουν να μπούμε εμεί και να κάνουμε ερωτήσεις για την προσωπική τους και την οικογενειακή ζωή. Από την άλλη υπάρχει ανάγκη να προστατευτούν αυτές οι πολύ ευάλωτε γυναίκες ε, που είναι κατά χιλιάδες στην Ευρώπη και εργάζονται σε σπίτια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ λεπτομερείς απαντήσεις για ζητήματα που έχουμε ακόμη να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας έχει λάβει πολλές πρωτοβουλίες σε σχέση με αυτό και θα δούμε τι θα γίνει και με την Γενική Συνέλευση Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας για το τελευταίο θέμα που αναφέρατε. Ε, δυστυχώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε άλλο αυτό το θέμα. Είναι η σκληρή ζωή της ε, κοινοβουλευτική μας επιτροπής που μας υποχρεώνει να σταματήσουμε εδώ τη σημερινή μας ανταλλαγή απόψεων. Όμως ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε και πάλι τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξής μας. Εξέταση τροπολογιών ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης που συντάσσουμε για την επί της ουσίας Επιτροπή Ήτρε για, την για, για, το θέμα αντιμέτωπης στο πρόβλημα της ασφάλειας των υπεράγριων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου. Ε, η συγγήτρια είμαι εγώ, 32 είναι οι τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί, εκ των οποίων 9 ε, τις έχω καταθέσει εγώ ίδια δεν πρόκειται δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγες είναι οι ε, τροπολογίες οι οποίες μας δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα. Έξι συμβιβαστικές τροπολογίες έχουν ε, δοθεί και στον σκιώδη εισηγητή, από τον οποίο δεν έχω λάβει παρατηρήσεις. Υποθέτω λοιπόν ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα και επομένως μπορούμε να τις ψηφίσουμε όπως τις έχω προτείνει. Για το σύνολο τώρα των ε, τροπολογιών, Κάποιες ζητούν ε, περισσότερες διευκρινήσεις ε, για τους χρόνους εργασίας στις πλατφόρμες των υπεράκτιων δραστηριοτήτων και λόγω του κινδύνου και λόγω της ιατρικής παρακολούθησης που χρειάζονται τέτοιου είδους δύσκολες συνθήκες εργασίας. Υπάρχει και μία ακόμη κατηγορία όσον αφορά την πληροφόρηση των ε, εργαζομένων για τις διαδικασίες ε, ε, ασφάλειας και για τους κινδύνους ε, στους οποίους εκτίθενται, όπως επίσης ε, και για τις, τους υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται σε πλατφόρμες τέτοιου είδους υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Ζητούμε λίγο μεγαλύτερη διαφάνεια των εκθέσεων παρακολούθησης και των ατυχημάτων που έχουν συμβεί, λίγο περισσότερη πληροφόρηση, γνωρίζουν περισσότερα οι αρμόδιες αρχές ε, καλύτερη εξέταση των ε, κινδύνων και των ενδεχομένων κινδύνων και τελευταία πτυχή ε, είναι το να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι στην αμοιβή του εργαζομένου. Αυτά ελπίζω ότι συνοψίζουν το πνεύμα των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Οπότε Υποθέτω ότι σας υπενθύμησα και το πνεύμα των συμβιβαστικών τροπολογιών. Ο κύριος Ορή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά σχόλια να κάνω. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι πολύ καλή και οι συμβαστικές τροπολογίες ε, θεωρώ ότι συνοψίζουν τις ε, θέσεις όλων συμπεριλαμβανομένων και των δικών μου. Άρα ε, το μόνο πρόβλημά μου είναι η συμβιβαστική πρόταση ΔΕΛΤΑ. Δεν μπορώ να τη δεχτώ. Η Λύση και εγώ κάναμε μια τροπολογία και οι δυο μας αυτό το οποίο θέλαμε είναι να υπάρχει μια αντί για να έχουμε μια μέγιστη εναρμόνιση, να έχουμε μια ελάχιστη εναρμόνιση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, εάν διατηρηθεί το κείμενο ως έχει, δηλαδή με μέγιστη εναρμόνιση, δεν θα συμφωνήσουμε. Προτιμούμε το αρχικό κείμενο. Ναι, αλλά το αρχικό κείμενο μιλούσε για μέγιστη εναρμόνιση. Τέλος πάνω, ο κύριος Κλάρκ και μετά η κυρία Λίνα. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν στην τροπολογία 6 που θα ψηφίσουμε αργότερα το απόγευμα λέει υπογραμμίζει ότι κάποια κράτη-μέλη ήδη έχουν εξαιρετικούς μηχανισμούς ασφαλείας σε σύγκριση με διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θα ψηφίσω υπέρ και θα έλεγα ότι πηγαίνει στην καρδιά της ασφάλειας των παράκτιων εγκαταστάσεων Πόσο μάλλον που ε, στοιχειοθετεί η βέλτιστη πρακτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω θα πρέπει να υιοθετούμε βέλτιστες πρακτικές από όπου και αν έρχονται. Αφού ισχύει αυτό, γιατί χρειάζονται γιατί χρειάζεται η σύνθετη αυτή καινούρια οδηγία, γιατί να μην υιοθετήσουμε τη βέλτιστη πρακτική, να κάνουμε τις τροποποιήσεις που πρέπει και να τελειώνουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επανεφεύρουμε τον τροχό εμείς εδώ. Δεύτερον, ε, από το πρωτότυπο κείμενο στην παράγραφο 7 καλεί τις εταιρείε που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες σε όλο τον κόσμο. Ε, είμαι, ακούγομαι κοινικός, αλλά κάποιες εταιρείε θα κάνουν μετεγκατάσταση και θα φύγουν από την Ευρώπη για να πάνε να εκμεταλλευτούν τα χαμηλότερα πρότυπα αλλού στον κόσμο για να συνεχίσουν τη δουλειά τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Και αν συμβεί αυτό το πράγμα, Βέβαια, θα πάρουν τις επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χάσουμε όλα τα εταιρικά κέρδη και τους φόρους. Δηλαδή, είναι σαν να πυροβολούμε το ίδιο μας το πόδι. Και δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα αυτή, δεν με ικανοποιεί. Ευχαριστώ, κυρία Λίν. Ε, συμφωνώ με τις ε, κυριότερες τροπολογίες ε, και τις συμβιβαστικές. Ε, η είμαι με απασχολεί λίγο γιατί έχω την τροπολογία 1, εγώ δική μου. Θα καταψηφίσω με την συμβιβαστική Α και θα πάμε στη δική μου τροπολογία 1. Στη Β έχω πάλι μια τροπολογία που την προτιμώ εγώ, δική μου. Την τροπολογία 4 θα καταψηφίσω με τη συμβιβαστική Β λοιπόν, ενώ θα ψηφίσω με υπέρ της τροπολογίας 40 αυτού. Υπάρχουν κάποια άλλα μικροπράγματα, πάντως γενικότερα η έκθεση είναι καλή και θα πρέπει να δουλέψουμε να, για να έχουμε κοινέ πρακτικές σε όλες τις λειτουργίες μας και επιχειρήσεις. Και είναι σημαντικό να γίνει αναφορά και στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε την υγεία και την ασφάλεια μέσα από ένα παγκόσμιο πρίσμα αρχίζοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά θα δουλέψουμε για να επιτύχουμε ε, συνολική συμφωνία για την υγεία και την ασφάλεια στις παράκτιες εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, θα απαντήσω στις ερωτήσεις και θα ξεκινήσω από τον κύριο Κλάρκ σε σχέση με το θέμα των βέλτιστων πρακτικών. Κοιτάξτε, κατά μία έννοια, ο στόχος αυτής της αναθεώρησης είναι να εμπνέεται κανείς από τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν. Οπότε νομίζω ότι λαμβάνεται υπόψη ε, η ανησυχία που εκφράσατε. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των ε, επιχειρήσεών μας στο εξωτερικό, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα των ίδιων μας των αντιφάσεων. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε ε, ως βίβλο την παγκό, της, ε, της, ε, του στόχου της χιλιετίας και μετά να πρέπει να δασκαλεύουμε τις επιχειρήσεις μας για το πώς θα φέρονται στο εξωτερικό. Τώρα, όσον αφορά το συμβιβασμό B, για τον οποίο μίλησαν, μίλησε η κυρία Λίνε και ο κύριος Ορή. Κοιτάξτε, εγώ τα είχα προσθέσει στην τροπολογία μου τις δικές σας ανησυχίες και διαπιστώνω ότι τώρα δεν είστε ικανοποιημένοι. Αν θέλετε, το end not minimum και όχι ελάχιστο να το διαγράψουμε και σε αυτή την περίπτωση θα σήμαινε μία ε, προσέγγιση που θα βασίζεται στην μέγιστη ε, δηλαδή αν θέλετε να, αλλάξουμε, να υπάρχει το μέγιστη εν προκειμένου. Θα ήθελα όμως ε, να σας υπενθυμίσω ε, τη σημασία του κειμένου αυτού. Αν δεν θέλουμε να έχουμε άριστες συνθήκες ε, εργασίας ε, και ε, αν δεν το θεωρούμε αυτό πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε ότι τα ανθρώπινα λάθη πολλές φορές προέρχονται από πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας στις πλατφόρμες αυτές υπεράκτιες και ξέρουμε ότι υπάρχει ήδη ιδιαίτερη ρύθμιση των συγκεκριμένων συνθήκων Βλέπετε όμως ότι η ελάχιστη αμέλεια μπορεί να έχει τεράστιες καταστροφικές συνέπειες. Οπότε πιστεύω ότι θα έπρεπε να ε, ζητήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, μέγιστη εναρμόνιση όπως είπα και προηγουμένως. Euh, αυτή είναι λοιπόν η πρόταση που σας κάνω και αν δεν θέλετε να τη δεχθείτε θα έχουμε ένα πρόβλημα γιατί οι τροπολογίες 4 και 5 δεν ε, μπορούν να θεωρηθούν ε, προσθήκες στη συμβιβαστική B. Όσον αφορά τη συμβιβαστική Α, πρέπει να πω ότι μου κάνετε εντύπωση, κυρία Λίνε, που δεν μπορείτε να το στηρίξετε, γιατί η τροπολογία σας 1 την έχω λάβει υπόψη όλοι στο τέλος της βιβαστικής A. Οπότε μου κάνει εντύπωση που δεν μπορείτε να υποστηρίξετε συγκεκριμένη ε, τροπολογία. Για τους λόγους σας εξήγησα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο παραπάνω μπορώ να κάνω. Είναι γεγονός ότι στην αρχή της ε, τροπολογίας ε, αναφέρομαι έχω συμπεριλάβει την τροπολογία 1, την οποία εσείς υποβάλατε, αλλά και την τροπολογία 2 του κυρίου Ορή όμως δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω μπορώ να κάνω από αυτό το οποίο έχω ήδη συμπεριλάβει στην συμβιβαστική α. Εγώ θα ήθελα λίγο περισσότερα πράγματα να συμπεριληφθούν. Για τις ασφαλιστικές εταιρείε μιλάω. Τότε κοιτάξτε. Ας κάνουμε τότε ξεχωριστή ψηφοφορία κυρία Λίνη, γιατί προφανώς έχετε πρόβλημα με την τροπολογία 3 του κυρίου Μπουλό. Αν καταψηφιστεί η συμβιβαστική Α που είναι πρώτη στον κατάλογο της ψηφοφορίας, τι προτείνετε τότε. Να μην αναφέρετε καθόλου το θέμα των ασφαλιστικών εταιριών. Κοιτάξτε, προτείνω ξεχωριστή ψηφοφορία. Ε, μου λένε ότι δεν γίνεται στη συγκεκριμένη επιτροπή για τέτοιου είδους θέματα. Κοιτάξτε, είναι ανόητος ο κανόνας. Ε, συγγνώμη, το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, je, Λοιπόν, ολοκληρώσω. Πιστεύω ότι η συμβιβαστική α θα μπορούσε να ε, ψηφιστεί ως έχει. Τώρα εντάξει, αν το ΕΛΚ διαφωνεί, αν ψηφίσει ό,τι θέλει και αν θέλετε, αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη δυσκολία με το τελευταίο τμήμα της συμβιβαστική α, εγώ προτείνω να, να συνεισφέρετε στη βελτίωση της διατύπωσης, αλλά νομίζω ότι είναι κρίμα να χαθεί αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, Ελπίζω να σας έπεισα για το πρόβλημα της ε, μέγιστης ενερμόνησης. Ο κύριος ορι Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Για την συμβαστική λύση Α δεν έχουμε πρόβλημα. Την ε, υποστηρίζουμε. Το Β, το Β τελικά είναι αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε και μας ε, δημιουργεί προβλήματα η, το μέγιστη, μέγιστη εναρμόνιση. Αυτό ε, ήθελα να πω και πριν. Δεν μας ενδιαφέρει το μέγιστη ή το ελάχιστη τέλος πάντων. Ε, ο επιθετικός προσδιορισμός μας ενοχλεί. Αν μείνει ως έχει το κείμενο, θα ψηφίσουμε την τροπολογία Λίνε και άλλων, την οποία υποστηρίζουμε. je vais rediscuter en coordinateur les conditions de vote des amendements de compromis. Euh, Mais pour l'instant. Αυτό το οποίο σας προτείνω είναι να αφήσουμε την έννοια της εναρμόνισης και να μιλήσουμε για common standards, based on common standards. Ή ή αλλιώς να παραμείνουν στο αρχικό κείμενο. Δέχεστε το common standards, να μιλήσουμε για common standards. you accept uh, uh, uh, to modify the compromise B and to Είπα να αλλάξουμε την ε, συμβαστική πρόταση ε, την, την ε, συμβαστική πρόταση Β και αντί να αναφέρουμε την μέγιστη ή την ελάχιστη εναρμόνιση να μιλάμε για common standards. Συμφωνείτε? Ωραία. Άρα τροποποιούμε με προφορική τροπολογία τη συμβαστική τροπολογία Β και αλλάζουμε το maximum ε, based on maximum or minimum harmonization με το common, ε, based on common standards. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και επομένως αύριο Α, όχι, όχι, σε λίγο θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση αυτή με βάση όλα αυτά τα οποία είπαμε. Περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης την ε, εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών για την έκθεση του κύριου Κόζα και που αφορά την κινητικότητα και την έμεξη των ατόμων με αναπηρίες. Ο κύριος Κόζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δουλέψαμε σκληρά και αρκετά οφείλω να ομολογήσω. Ευχαριστώ για την συνεργασία τους ε, σκιώδης εισηγητές και από τις 28 συμβαστικές τροπολογίες μία μόνο παραμένει ακόμα σε κρεμότητα. Και για αυτήν τη συμβαστική τροπολογία θα ήθελα να... Μάλλον τρεις τροπολογίες είναι ε, συμβαστικές τροπολογίες που παραμένουν σε κρεμότητα. Ε, η πρώτη συμβαστική τροπολογία είναι η γάμα για την οποία ήθελα να σας μιλήσω. Εδώ να σας πω ότι οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν. Α, υπάρχει ένα πρόβλημα με την γερμανική διερμηνία. Τέλος πάντων, κύριε Σεγητά, έχετε το λόγο ξανά. Λοιπόν, θα επαναλάβω από την αρχή αυτά που είπα. Σας είπα ότι δουλέψαμε σκληρά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συγητές για τη συνεργασία τους. Να σας πω ότι από τις 28 συμβαστικές, τροπο, μάλλον 28 συμβαστικές τροπολογίες ε, ε, είναι μπροστά μας, εκ των οποίων μία και μόνο ε, παραμένει σε κρεμότητα. Λοιπόν, να σας μιλήσω για τρεις, συμβαστικές, για τρεις τροπολογίες και για τις οποίες θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Καταρχάς έχουμε τη συμβαστική τροπολογία Γ. Να δούμε, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, να σας πω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν με την συμβαστική αυτή λύση. Η πιο μεγάλη ένωση οργάνωσης ε, ε, των ατόμων με, με αναπηρία είναι αντίθετη όμως με την, ε, ε, με την τροπολογία αυτή, γι' αυτό θεώρησα σκόπιμο να το αναφέρω. Μιλάμε για την ίδρυση μιας οργάνωσης που θα παρακολουθεί την ζωή των ατόμων με αναπηρία. Στο αρχικό κείμενο αναφέραμε τον όρο κοινότητα. Αλλά αυτός ο όρος είναι ήδη, χρησιμο... ήδη χρησιμοποιείται. Άρα δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς. Ε, προτείνουμε τον, επίσης έναν άλλον όρο που προτείνουμε εμείς είναι ο όρος πλατφόρμα. Όμως υπάρχει και άλλη μια πρόταση. Αντί να μιλήσουμε για πλατφόρμα, να, μιλάσουμε, να μιλήσουμε για πυρήνα, για board, για συμβούλιο. Να σας πω ότι, με... ότι έχουμε και μία δική μου τροπολογία εδώ για την δημιουργία του συμβουλίου αυτού χρειάζεται μία διαθεσμική, αν θέλετε, συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, Έχουμε την συμβαστική τροπολογία Π. Εδώ οι απόψεις συγκλίνουν. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω στο σημείο αυτό. Να σας πω επίσης ότι η συζήτηση γίνεται για να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της προστατευμένης απασχόλησης όσον αφορά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Η επόμενη συμβαστική τροπολογία, η Q, αφορά την οριζόντια οδηγία. Φύλλο, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία είναι μια, πρόκειται για μια οδηγία που είναι ανεξάρτητη τέλο πάντων και αποφορά τα θέματα αυτά. Εγώ προσπάθησα να κάνω μια να υποβάλω μια τροπολογία και υποβάλω μια τροπολογία και να σας πω ότι οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι υπέβαλαν μια άλλη συμβαστική τροπολογία η οποία υπάρχει στον κατάλογο ψηφοφοριών Το ΕΛΚ δεν την υποστηρίζει την ε, πρόταση αυτή, την τροπολογία αυτή. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προηγούμενη συζήτηση ε, και ε, που ακούσαμε την άποψη της Προέδρου. Είπε ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ξεχωριστά την συμβαστική τροπολογία. Να σας πω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μέλη τα οποία θα, θα ήθελαν να γίνει κάτι τέτοιο, διότι θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε σε δύο τμήματα την συμβαστική τροπολογία. Τέλος πάντων, πέραν τούτου νομίζω ότι όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες ε, όλοι συμφωνούν. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια, ότι όταν ενταχθούν οι τροπολογίες αυτές στην έκθεση, η έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα καλύπτει το σύνολο της ζωής των ατόμων με αναπηρία. Και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το περιμένω αυτό. Ευχαριστώ. Δυστυχώς, κύριε εισηγητέ, ε, με επανέφεραν στην τάξη δεν έχω δικαίωμα να ζητήσω ξεχωριστή ψηφοφορία ε, όσον αφορά τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε πριν, στη δική μου έκθεση δεν θα μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Κυρία Μπλίνκεβιτς και μετά η κυρία Λίνε. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να πω ότι οι διαπραγματεύσεις ε, επί των συμβιβαστικών τροπολογιών δεν είναι εύκολες, κάποιες φορές δυσκολεύουν και πάρα πολύ και περιπλέκονται. Καμιά φορά οι προτάσεις από τα άλλα κόμματα δεν είναι κατανοητές αμέσως, όμως χαίρομαι που βλέπω το τελικό αποτέλεσμα και Είμαι ευτυχής διότι ο εισηγητής κύριος κόσα συμπεριέλαβε κάποιες προτάσεις των σοσιαλιστών δημοκρατών, φιλελευθέρων πρασίνων και έχουμε συμφωνήσει επί ορισμένων συμβιβαστικών τροπολογιών, παρόλο που χτες είχαμε διεστάμενες απόψεις. Άρα χαιρόμαστε πολύ. Τώρα διότι Καμία ομάδα δεν θέλει να επιδεινωθεί η κατάσταση αυτών των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με τη συμβιβαστική Q, ε, εμείς μιλάμε εδώ για το Κοινοβούλιο που θα προσελκύσει την προσοχή των κρατών μελών στη σημασία του θέματος των διακρίσεων και της οδηγίας για τις διακρίσεις, την διακριτική μεταχείριση. Αν λέμε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρίες και να τους φροντίσουμε όπως τους αξίζει. Σήμερα το πρωί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μας ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουγγρική Προεδρία σχετικά με την κατάσταση για την οδηγία αυτή ακριβώς. Και ο εισηγητής Κώσα ήταν παρόν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στην πρωινή της συνεδρίαση και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Ουγγρική Προεδρία ε, παρέσχε πληροφορίες και είπε δηλαδή ότι κατά τη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας της ε, επικεντρώθηκε στο θέμα ε, των ανθρώπων με αναπηρίες. Δουλεύουν πάνω στην οδηγία για τις αναπηρίες και η Ουγγρική Προεδρία προσπάθησε να εντάξει όλα τα θέματα στα πλαίσια αυτής της οδηγίας και θα ήταν πολύ καλή ιδέα θεωρώ να υποστηρίξουμε τη συμβιβαστική πρόταση σχετικά με την ανάγκη ταχύτερης εξέλιξης της οδηγίας για τις διακρίσεις και την, ε, τις Και επειδή δεν βρέθηκε λύση κοινή, μαζί με τον εισηγητή προτείναμε και οι σοσιαλιστές δημοκράτες και οι πράσινοι είπαμε να υποβάλλουμε συμβιβαστική τροπολογία Πρώτον, να γίνει κατανοητό ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ τα απαραίτητα ε, ε, κονδύλια, είτε ζούμε σε εποχή οικονομικής κρίσης είτε όχι, ποτέ δεν θα φτάσουν τα ε, κονδύλια. Και αυτό που βλέπουμε στα κρατη σε κάποια κράτη-μέλη είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης για να ασχοληθούν με τα θέματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Οπότε εδώ χρειάζεται πολιτική βούληξη να συμφωνήσουμε με τις ε, συμβαστικές. Η κυρία Αλίν, ευχαριστώ πολύ γιατί Άνταμ έλαβε υπόψη σου πολλές προτάσεις. Προτάσεις μας έχουμε τώρα ένα κείμενο που εν πολλής είναι αποδεκτό στην πλειοψηφία των ε, συναδέλφων. Βέβαια ε, μένουν κάποιοι τομείς που πρέπει να συζητηθούν, αλλά πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση με το κείμενο, γιατί αυτό το δουλέψαμε πολύ καιρό και τώρα έχουμε τη σωστή προσθέγγιση με βάση τα δικαιώματα και όχι την αναπηρία. Τώρα για την τροπολογία τη συμβαστική αν θα μιλήσουμε για πλατφόρμα, για συμβούλιο, για επιτροπή ε, αναπηρίας, ε, ε, θα θέλαμε να μιλήσουμε για επιτροπή, λένε μερικοί. Τώρα, εγώ είμαι ανοιχτή πλατφόρμα, συμβούλιο, επιτροπή. Δεν με νοιάζει πώς θα τη λέμε. Αρκεί να κάνει το σωστό. Να παρακολουθεί δηλαδή τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν με νοιάζει πώς θα το πούμε. Έτσι λοιπόν, ε, αν μπορούμε να ε, έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας, ε, εγώ θα συμφωνήσω σε οτιδήποτε. Οτιδήποτε και να πούμε στη συμβαστική C. Τώρα για τη συμβαστική P, Εφιστώ την προσοχή σας σε ορισμένα προβλήματα που εξακολουθώ να έχω με τη συμβαστική π, π, συμβαστική τροπολογία π. Ε, έγιναν συζητήσεις και με τους ε, πράσινους και με τους σοσιαλιστές δημοκράτες για αυτό το θέμα και με τη EDF ε, και με άλλες οργανώσεις ανθρώπων με αναπηρίες για να έχουμε μια συμβαστική λύση που θα καλύψει πολλά από αυτά που αναφέρονται στις τροπολογίες αλλά να τα ξαναδούμε και να έχουμε μια συνοχή στις τροπολογίες γιατί έτσι όπως είναι τώρα διατυπωμένη η τροπολογία αναφερόμεθα σε προστατευόμενα εργαστήρια στην αρχή και μετά ε, τα λέμε πολύ και στη μέση της έκθεσης. Επίσης καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τα προεκπροστατευόμενα εργαστήρια ω μέσον και να συνάψουν συμβάσεις ε, τα οποία θα, ε, ανταποκρίνουν, θα λαμβάνουν υπόψη την επιμέρους αναπηρία. Και με ε, βάση μια διαδικασία κατάρτισης πολύ υποστήριξη στο αρχικό στάδιο. Στην αρχή δεν το θέλαμε εμείς αυτό. Σε ορισμένα κράτη-μέλη υπήρχε η διαδικασία αυτή. Ε, άλλοι είχαν σύστημα ποσοστώσεων, το οποίο μετά ε, δεν το ε, εφάρμοζαν τόσο πολύ. Τώρα, για τα προστατευόμενα εργαστήρια δεν είμαι κατά, αλλά είναι και ένα εφαλτήριο, αν θέλετε, για την απασχόληση, δεν αντικαθιστά λέμε καλή τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τα προστατευόμενα εργαστήρια. Ε, το τονίζουμε πολύ το πρώτο μέρος και μετά στο μέσον λέμε, κάνουμε το αντίθετο. Γι' αυτό σας έστειλα μια διαφορετική συμβιβαστική και οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι την εξέτασαν ε, και είχα απάντηση από τους πράσινους και είπαν ότι το υποστηρίζουν. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση αφού εξετάσετε και εσείς αυτή την τροπολογία, γιατί οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι συμφωνούν. Για τη συμβαστική Q νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, λυπάμαι που δεν θεωρήσατε πρέπει να καταθέσετε τις τροπολογίες πρασίνων και σοσιαλιστών, δεν ήμουν εγώ να υποβάλλω, για την οδηγία για τις αναπηρίες που είναι τόσο σημαντικό θέμα. Χαίρομαι διότι προχώρησε η συμβαστική Q. Ακόμα και σε αυτό το όψιμο στάδιο, ελπίζω να συμφωνήσετε στην τροπολογία τη συμβαστική Q, γιατί κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των οργανώσεων των, για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, υπάρχει σύμφωνη γνώμη ότι είναι πολύ σημαντικό η οδηγία αυτή να αξιοποιηθεί για να προχωρήσουμε στο θέμα αναπηρίες. Ξέρω και το ε, EDF, e το European Disability ε, φόρουμ συμφωνεί και άλλοι και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε με τη συμβαστική Q όταν θα καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος ψηφοφοριών. Κάποια κράτη-μέλη είναι κατά, αλλά μου φαίνεται ότι το κυρίο σώμα του Κοινοβουλίου είναι υπέρ. Ο κύριος Τόμας Μαν και μετά η κυρία Σρότερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Άνταμ Κόζα για την εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ ώστε να εξεύρουμε συμβιβαστικές λύσεις και αυτό είναι σημαντικό μήνυμα. Όχι μόνο για τις οργανώσεις των αναπήρων αλλά και τους πολλούς που περιμένουν από εμά συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όχι να μόνο θεωρητικολογίες. Είναι σημαντικό μήνυμα και αν δω, δω που πέτυχαν οι υπεύθυνοι των ομάδων ισχυώδης, πραγματικά κάναμε τεράστια βήματα μπροστά. Τώρα, για την τροπολογία C, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια φόρμουλα, ε, όπως ε, πρότεινε ο Άνταμ Κόζα, κομίτη, επιτροπή. Είναι σημαντικό. Οι οργανώσεις των αναπήρων θέλουν να ε, υιοθετήσουν μια τέτοια θέση. Θέλουν μια τέτοια θέση. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, πιστεύω. Τώρα, ε, κάποια προβλήματα υπάρχουν στην Q. Η κυρία Λίν ε, αναφέρθηκε στο θέμα, μιλήσαμε και για τις διακρίσεις και αν χρειάζεται νέα νομοθεσία. Αν δούμε το δεύτερο μέρος, συζητή από την Κομισιόν μέχρι το People with Disability, ε, δεν είναι ξεκάθαρο τι θέλουμε. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές εδώ μεταξύ των πολιτικών ομάδων μας. Όλοι θέλουν να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα αυτών. Όλοι θέλουν η νομοθεσία κατά των διακρίσεων να συμβάλλει ε, στην άρση των κοινωνικών εμποδίων. Όλοι θέλουμε να καταφέρουμε τα άτομα με αναπηρίες να είναι αποδεκτά και θέλουμε να υπάρχει σχετική νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Στο πρώτο μέρος ε, λέει πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια νέα οδηγία. Εδώ διατυπώνονται οι διαφορές, ε, εδώ ε, υπάρχουν διαφορές. Η κυρία Ελίν αναφέρθηκε στην συμβιβαστική πι και είπε ότι ανέπτυξε μια εναλλακτική σε ένα κομμάτι του. Αν τα καταφέρουμε στο π να επιφέρουμε αλλαγές, τότε θα πρέπει να δούμε μήπως μπορούμε και στο Q. Κουνάει το κεφάλι γραμματεία. Δεν μπορούμε δηλαδή. Δεν μπορούμε στη... Α, λέτε, δεν μπορούμε να δεχτούμε σε μια συμβιβαστική το πρώτο κομμάτι και όχι το δεύτερο. Αλλά αν καταλήξουμε όλοι ότι θα έχουμε ένα έργο που θα, μας, θα το δουλέψουμε όλοι, ε, αξίζει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, αν σε αυτή την περίπτωση στο Q, στο πρώτο τμήμα δεν ε, επιτύχουμε σύμφωνη γνώμη και ούτε με τον εισηγητή, αλλά συμφωνήσουμε στο δεύτερο κομμάτι, θα ήταν σόφρον και έξυπνο να πούμε, για να δούμε να τροποποιηθεί η Q και να μείνει το δεύτερο κομμάτι. Δηλαδή, ε, μπορούμε και το τυπικό θέμα να το λύσουμε. Γενικά νομίζω ότι ε, ενσωματώσαμε πολλές εξαιρετικές προτάσεις μετά από πολλές επαφές με τις οργανώσεις των αναπήρων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μας ε, βοηθάει να προχωρήσουμε. Η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας ελπίζω να μην αντιμετωπιστεί όπως κι άλλες που περιθωριακά εξετάζονται. Δεν επιτρέπεται αυτό, πρέπει να γίνει σοβαρή και σημαντική συζήτηση. Και πολλοί από την Επιτροπή μας δούλεψαν πολύ και ενδιαφέρονται για μια επιτυχία που θα είναι επιτυχία όλων μας. Πάλι ευχαριστώ Άνταμ και ευχαριστώ και όλους που δούλεψαν με τόσο θετικό πνεύμα πάνω σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να ενώσω τη φωνή μου ε, σε εκείνοι αυτών που έδειξαν ε, βούληση για συνεργασία, γιατί αυτό βελτίωσε τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες και σύμφωνα με το τελευταίο κείμενο που έχω εγώ υπάρχουν τρεις συμβιβαστικές που δεν μπορούμε να στηρίξουμε και ένα τέταρτο πρόβλημα που το τέταρτο είναι η οδηγία κατά των διακρίσεων. Θα μιλήσω και γι' αυτό, αλλά για τις τρεις συμβιβαστικέ θα έλεγα ότι οι πράσινοι συμφωνούν με την α και την ε μου φαίνεται η δεύτερη, όχι όμως με την π, εκεί ε, θα στηρίξω με την πρόταση της ε, ε, κυρίας Λίν για τα προστατευόμενα εργαστήρια, sheltered workshops, το είπαν και οι ειδικοί, ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι το σημαντικό θέμα. Αυτό δεν αποκλείει να ε, περάσουν και σε προστατευόμενα εργαστήρια και μετά στην ε, αγορά εργασίας να αξιοποιήσουν αυτά τα εργαστήρια, αλλά εδώ πρέπει να είμαστε μαξιμαλιστές στα αιτήματά μας. Είναι σημαντικό αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι ξεκάθαρη άλλωστε. Μιλάει για ελεύθερη πρόσβαση στις αντίστοιχε οδηγίες κατά των διακρίσεων. Το θέμα πώς θα καταλήξουμε εκεί αυτό ε, θα το ρυθμίσουν τα κράτη-μέλη αλλά θα πρέπει να τηρηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι' αυτό στηρίζουμε την πρόταση της Λισλίν και θα πρέπει να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σχετικά με το ΠΕ. Ακούσαμε και άλλα πράγματα. Είμαστε διατεθειμένοι να προσεγγίσουμε ένα στον άλλον, αλλά καταρχήν στηρίζουμε την πρόταση της Λιν. Τώρα, για την οδηγία κατά των διακρίσεων. Εκπλήσωμε που ο εισηγητής σε κάποια άλλα σημεία της έκθεσης του θέτει νομοθετικά αιτήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάει για τις διάφορες γλώσσες που πρέπει να είναι ορατές. Ε, εδώ πρόκειται για σχεδιασμό έξυπνων τηλεφώνων κλπ. Απόλυτα θεμητό. Είναι ένα ευρύ αίτημα. Και υπάρχουν εδώ νομοθετικές ε, προδιαγραφές. Αλλά όταν πρόκειται για νομοθετικές προτάσεις για την οδηγία κατά των διακρίσεων, ε, δεν αναφέρει τις αντιρρήσεις κάποιων συναδέλφων. Το ξέρουμε αυτό. Όταν προσπαθήσαμε να τα βρούμε κατά την πρώτη ανάγνωση στην οδηγία κατά των διακρίσεων. Ένα κράτος ήθελε να μπλοκάρει την υπόθεση και μετά κάποιοι βουλευτές καταψήφισαν. Δικαίωμά θα μου πείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ο εισηγητής εν προκειμένου ακολουθεί εκείνους και δεν έχει δική του θέση είναι πολύ σημαντικό να κατησχύσει εδώ η οδηγία κατά των διακρίσεων. Θα ε, πρέπει να δώσουμε πράσινο φως στην εξέλιξη αυτής της οδηγίας. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θα σκεφτούμε και εμείς ανάλογα αν θα υποστηρίξουμε ή όχι. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Φιγκουερέιντο. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω τη δουλειά των, ε, του εισηγητή μας. Ήταν, ε, επέδειξε πολύ ανοιχτό πνεύμα όσον αφορά τις απόψεις των διαφόρων συναδέλφων. Μόνο δύο-τρία ζητήματα θα ήθελα να τονίσω. Καταρχάς, η τροπολογία C. Το θέμα της πλατφόρμας. Το θέμα του ορισμού δεν είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό, νομίζω. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα είναι αποδεκτό από όλους ε, και από τους οργανισμούς, από τις οργανώσεις αναπήρων, γιατί δεν ε, νομίζω ότι χρειάζεται να δημιουργούμε θέμα εδώ ή να δημιουργηθεί πρόβλημα με τις οργανώσεις των αναπήρων. Δεύτερη παρατήρηση, ποσοστώσεις. ένα ζήτημα που συνεχώς ανακύπτει. Και η κυρία Λίνε και άλλοι που είναι πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουν ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητούμε πολύ συχνά. Ναι ή όχι στις ποσοστώσεις. Στον τομέα των αναπηριών είναι κάτι που δημιουργεί πάντοτε έντονες συζητήσεις. Εμείς θέλουμε να προβληματιστούμε επί του θέματος αυτού, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν αναπηρίες, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα απασχολησιμότητας. Υπάρχει πάντοτε μια διακριτική ε, μια τάση διακριτική μεταχείρισης και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό είμαστε λοιπόν αρκετά ανοιχτοί Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά δημιουργεί έντονες συζητήσεις, άλλοι θέλουν ποσοστώσεις, άλλοι όχι και γνωρίζουμε ότι το θέμα είναι ευαίσθητο. Και θα ήθελα να σας πω ολοκληρώνοντας ότι παρά το ανοιχτό πνεύμα που υπάρχει, είναι κρίμα που δεν έχει ο εισηγητής μία ακόμη πιο ανοιχτή ε, θέση που θα μπορούσε να συμπεριλάβει την προάσπιση της ύπαρξης ενός ελάχιστου μισθού. Είναι κάτι το οποίο είχαμε αποδεχθεί όταν ήμουν εγώ ε, εισηγήτρια για το θέμα αυτό του ελάχιστου, της ελάχιστης αμοιβή. Δεν ε, υπερασπίζομαι ένα ενιαίο ελάχιστο μισθό, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε κάπως να ανακουφίσουμε τη φτώχεια και είναι ένα ζήτημα θεμελιώδες νομίζω. Γιατί αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη μια συγκεκριμένη υποστήριξη, επιπλέον υποστήριξη μέσω μέτρων καταπολέμησης της φτώχειας, τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι με αναπηρίες, αυτοί είναι οι άνθρωποι που μερικές φορές είναι αντικείμενο διπλής και τριπλής διακριτικής μεταχείρισης. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε, κατά τη γνώμη μου, να συμπεριλάβουμε τη σχετική τροπολογία που μιλάει για αυτό το θέμα. Θέλει... Θέλετε να επανέλθετε σε ένα-δύο από τα σημεία τα οποία ακούστηκαν. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν. Νομίζω ότι οι λύσεις που επιλέξαμε είναι καλές. Επίσης, να σας πω ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες έχουν γίνει δεκτές από το σύνολο των πολιτικών ομάδων, εκτός από μία τροπολογία βέβαια. Άρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αν θέλετε, είναι υπέρ των συμβιβαστικών τροπολογιών. Τώρα βέβαια υπάρχουν οι τρεις αυτές οι βασικές τροπολογίες, P, Q και C, που θα πρέπει να ε, καταβληθεί μια προσπάθεια για να βρούμε έναν κοινό παρονομαστή. Λοιπόν, για το C να σας πω ότι δεν συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι το όνομα δεν έχει σημασία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι οι αρμοδιότητες. Τώρα, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον, και αυτό που είναι το σημαντικό είναι το κατά πόσον αυτές οι τρεις, ε, οι, αυτός ο οργανισμός αν θέλετε θα τύχει της... Ε, στην αρχική μου πρόταση έλεγα ότι φτάνουμε κοντά σε μια συμφωνία. Υπάρχουν τρεις προτάσεις δική μου, της κυρίας Λίν και τρίτον μια πρόταση των σοσιαλιστών. Αυτές οι τρεις προτάσεις, ωστόσο, βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια τη σημερινή ημέρα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα την υποστηρίξουν όλε οι πολιτικέ ομάδε σε σχέση με την τροπολογία που για τους ε, α, βαρύκους ή τους ε, με προβλήματα στην ακοή ανθρώπους. Ε, σε σχέση με τον συμβιβασμό, ελπίζω ότι θα υπάρξει υποστήριξη από πλευρά του Δεν έχω εγκαταλείψει την προσπάθεια. Θα καταλήξουμε, ελπίζω, σε ένα συμβιβασμό. Επίσης σε σχέση με την πρόταση του κυρίου Μαν που προτείνει την επιλογή μιας άλλης επίλυσης. Θα προβληματιστώ σε σχέση με αυτό και θα το δω. Θα έρθω σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές στο υπόλοιπο της ημέρας να δω τι μπορεί να γίνει. Είδα ότι υπάρχει μια τροπολογία Y, Y ελληνικό Y, που θα ε, αναφερόταν στο τρέχον έτος ε, και που αφορά ένα ε, πακέτο το οποίο ε, εμποδίων που πρέπει να, ε, προσκομμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ίσως με την επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε θα πρέπει να δούμε αυτή την προοπτική. Επίσης έχουμε και ένα άλλο σχόλιο το οποίο έγινε σε σχέση με τον ελάχιστο μισθό. Δεν θα ήθελα να υπησέλθω τώρα σε υπερβολικές λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Όχι επειδή δεν θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό, όχι, αλλά επειδή δεν θα ήθελα να επεκτείνω υπερβολικά το πλαίσιο της έκθεσης. Θα ήθελα να το περιορίσω, να το αναφέρω μόνο στο πλαίσιο των ρεαλιστικών δυνατοτήτων και λύσεων ως προοπτικών. Και τέλος για το σύστημα ποσοστώσεων σε σχέση με τις ποσοστώσεις. Θα ήθελα να πω ότι οι απόψεις είναι διαφορετικές και παρεκκλίνουν εγώ ως άτομο με μειονεξία, με ειδικέ ανάγκες και εδώ και τόσα χρόνια που προσπαθώ να ενταχθώ όσον αφορά τα προβλήματά μου, μπορώ να σας πω ότι η νομοθεσία δεν είναι αποτελεσματική. Το σύστημα των ποσοστώσεων σήμερα, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίο. Μακροπρόθεσμα, εντάξει, συμφωνώ να εξαλειφθεί, να πάψει να υφίσταται. Σήμερα όμως όχι. Είναι ανάγκη να υπάρχει ιδιαίτερα για την κεντρική Ευρώπη, είναι σημαντικό να αυξηθεί η απασχόληση των ατόμων με ειδικέ ανάγκε και αυτό μόνο μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύστημα ποσοστώσεων που θα μπορεί να λειτουργήσει. Με αυτά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συνένεση. Ευχαριστώ και πάλι για τι παρεμβάσει σα και ελπίζω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα σε σχέση με την ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ δεν θα είμαι κατά διάρκεια τη ψηφοφορία, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά οι αντιπρόεδροί μα. Πάμε στο σημείο 6 τώρα, όπου θα εξετάσουμε τι 12 συμβαστικέ ε, τροπολογίε που προτείνει ο κύριο Ουγγουρεάνου για την προώθηση ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ισηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε φτάσαμε στην τελική εκδοχή των συμβαστικών τροπολογιών. Ε, τις υποστηρίζουν πρακτικά όλες οι πολιτικές ομάδες και αυτό, κυρία Πρόεδρε, ε, οφείλεται στο γεγονός ότι οι συμβαστικές τροπολογίες συνδυάζουν ε, διάφορες απόψεις του πολιτικού φάσματος, αλλά και γιατί όλοι δέχονται την, τον θετικό χαρακτήρα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Υπάρχουν όμως και κάποιες απόψεις ε, που θεωρούν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων εργαζομένων ε, και οι πολλοί θεωρούν ότι η άρση αυτών των εμποδίων δεν αποτελεί ε, πανάκια δεν είναι μια πανευρωπαϊκή λύση αυτό. Και αυτό είναι ένα γεγονός, κυρία Πρόεδρε. Έχουν γίνει μελέτες που αποδεικνύουν ότι η κινητικότητα δουλεύει και η πιο πρόσφατη ιστορία μας έδειξε ότι δεν, υπήρχε, δεν είχαμε επαναστάσεις, ε, πολλέ, πόλεμοι, ε, λόγω της ε, του φόβου για την ε, ε, άφηξη των Ανατολικοευρωπαίων. Ίσα ίσα σε ανάπτυξη οδήγησε η άφηξη αυτή. Γι' αυτό ακριβώς κυρία Πρόεδρε καταλήξαμε σε αυτή την συμφωνία με όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Αυτά. Ευχαριστώ η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ και εγώ θα είμαι σύντομη. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του συνεργασία. Για τη συμβιβαστική ΣΥ θα ήθελα να μιλήσω. Θα την υποστηρίξουμε. Απλώς υπάρχει ένα σημείο που λέει ότι η ίση αμοιβή για την ε, ίδια εργασία στον ίδιο χώρο ε, λαμβάνεται υπόψη από κοινού με το θέμα της ισότητας των φύλων. Είχαμε κάποιο πρόβλημα με αυτό Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με τους προσωρινά εργαζομένους. Ε, μερικές φορές μάλιστα αυτοί πληρώνονται περισσότερο. Είναι κάτι που συμβαίνει στην Ιρλανδία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επί της γενικής αρχής μπορούμε να υποστηρίξουμε τη συμβιβαστική αφιτροπολογία. Ήθελα απλώς να κάνω το σχόλιο ότι υπάρχει το ζήτημα των προσωρινά εργαζομένων. Ε, δεν έχουμε πάρα πολύ χώρο, οπότε, χρόνο, οπότε δεν θα επιμείνω στα υπόλοιπά μου σχόλια. Κυρία Μπλινκεβίτσιούτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Γκουρεάνου, για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε μαζί του, για τη σκληρή δουλειά του κατά την προετοιμασία των συμβιβαστικών τροπολογιών. Ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, όμως στο τέλος τα καταφέραμε. Καταφέραμε να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα που βλέπετε και η ομάδα μας θα υποστηρίξει τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κι εγώ κάτι. θεωρώ ότι είναι καλό να πούμε ότι θα μας δώσει μια μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταλάβουμε τι έγινε ε, σε σχέση με την ελεύθερη διακίνηση, τι διαφορές είναι σημαντικό γιατί ορισμένοι φοβούνται ότι η ελεύθερη διακίνηση ε, θα οδηγήσει σε πλήρη αλλαγή. Όλα αυτά όμως δεν έγιναν, οι φόβοι δεν επαληθεύτηκαν. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό και σημαντικό είναι να έχουμε περισσότερα στοιχεία, περισσότερες τάσεις, ε, συσχετισμούς και να πούμε με βάση ε, έγκυρα στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λόγο για να μειωθούν οι φόβοι σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτό θα είναι μια καλή βάση. Υπάρχουν, ε, υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση σε κάποια κράτη-μέλη, ε, κάποιοι άλλοι φόβοι και μέτρα σχετικοποιήθηκαν γιατί πολλοί κατάλαβαν ότι είναι πολύτιμο αγαθό η ελεύθερη διακίνηση. Ε, αν ε, συμφωνήσουμε σε αυτό το γενικότερο πνεύμα θα μπορέσουμε να, έχουμε, να ψηφίσουμε καλή έκθεση και καλές συμβασικές τροπολογίες αύριο. Κύριε Σιγητά, μετά από όλους αυτούς επένους θέλετε να ξαναπάρετε το λόγο. Ναι, πολύ σύντομα δεν θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο. Καταλαβαίνω ότι είναι θεμητές οι ανησυχίες ε, που ε, αναφέρθηκαν. Νομίζω ότι μπορούμε ούτως ή άλλως να συνεργαστούμε και να ζητήσουμε μία μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γνωρίζουμε βέβαια για ποιο λόγο δεν έγινε η μελέτη ως τώρα, αλλά οι μελέτες είναι πάντα χρήσιμες. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την έκθεσή σας αύριο. Μας μένει ένα τελευταίο σημείο πριν από την ε, ψηφοφορία που είναι οι συμβιβαστικές τροπολογίες ε, της έκθεσης κυρίας Μπάουερ ε, για την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων για την απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Κυρία Μπάουερ, έχετε το λόγο. Thank you so much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την ειλικρίνεια των σκιωδών, οι οποίοι τόσες πολλές συμβιβαστικές ε, υπέβαλαν. Έχουμε 11 συμβιβαστικές μπροστά μας. Να αναφερθώ στην συμβιβαστική J, απεσύρθη η λέξη large, μεγάλες. Αυτή είναι μια σύντομη διευκρίνηση τώρα. Η διατύπωση είναι ε, λυπάται διότι τα κοντήλια δεν χρησιμοποιούνται. Ε, αυτό λόγω μακρών διοικητικών διαδικασιών κλπ. Αυτά είναι χρήματα που υπήρχαν από προηγούμενες προγραμματικές ε, περιόδους ε, και με δυσκολία χρησιμοποιούνται. Δεν... Καλό είναι να μην, χρησιμοποιήσουμε, αυτή τη φρασιολογία ότι πολλά χρήματα μένουν αδιάθετα, οι πιστώσεις δηλαδή χρησιμοποιούνται. Να έχετε υπόψη σας ότι η λέξη large έχει φύγει. Τώρα για τις νέες εξελίξεις έχουμε νέα συμβιβαστική, 12η επί τη βάση της τροπολογίας 46. Σήμερα καταλήξαμε εκεί και θα σας δοθεί και σε εσά αύριο. Με την εξής διατύπωση καλή τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ε, επαγγελματικά ε, shops για να βοηθήσουν στην εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής και με τις τοπικές αρχές και με τους πολίτες της Ένωσης. Αυτή είναι η επόμενη συμβιβαστική που θα την πάρετε γραπτός για να τη δείτε. Ένα ακόμα θέμα ε, θα ήθελα να πω στους συναδέλφους σχετικά με τον κατάλογο ψηφοφορίας. Αν εφαρμόσουμε τον κανόνα 161 από τη γραμματεία, αν εφαρμοστεί ο κανόνας αυτός, ε, θα δούμε ότι υπάρχουν κάποιες εκρεμείς τροπολογίες πριν από τις συμβιβαστικές. Μερικές από αυτές ε, είναι απόλυτα εντάξει, αλλά αναφέρονται εν μέρη σε διαφορετικά πράγματα, οπότε δεν εντάχθηκαν στην ε, γνωμοδότηση. Για παράδειγμα, έχουμε την παράγραφο 1 και την τροπολογία 5 της κυρίας Κώστα. Κανένα πρόβλημα με το περιεχόμενο, συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν εστιάζει στο θέμα μας, εστιάζει στη στρατηγική 2020. Αν αυτές οι τροπολογίες εγκριθούν, θα καταπέσουν οι συμβιβαστικές όμως και το αποτέλεσμα είναι, θα είναι αβέβαιο. Προσέξτε λοιπόν, εμείς έχουμε καταλήξει σε ε, ευρείες συμβιβαστικές με διάφορες πολιτικές ομάδες και σας καλώ να υποστηρίξετε και να υπερψηφίσετε τις συμβιβαστικές και όχι αυτές τις τροπολογίες οι οποίες επί της ουσίας όπως σας είπα πολλές φορές είναι πολύ εντάξει αλλά αναφέρονται σε άλλα πράγματα και αλλάζουν άρδιν το κείμενο. Είναι κανείς άλλος να πάρει το λόγο? Μάλλον όχι, οπότε θα ψηφίσουμε επί τη βάση των συστάσεων της εισηγήτριάς μας, επί του συνόλου των ε, συμβιβαστικών τροπολογιών και των υπολείπων τροπολογιών αύριο. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία μας και ξεκινούμε με το 8 με τη γνωμοδότηση για το πρόβλημα της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων ε, εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου για την Επιτροπή Ήτρε για την παράγραφο 1 συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 συμβιβαστική β. Όπως θα θυμάστε, αλλάξαμε το κείμενο, έχουμε προφορική τροπολογία, ο, έχουμε ε, όχι μέγιστη εναρμόνιση, αλλά common standards, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 6, μαν, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 το μασμάν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική σε παράγραφος 4 υπέρ. Συγγνώμη λέει η πρόεδρος. Παράγραφος 3. Ξέχασα την τροπολογία από το της κυρία Στάιντρουκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά πάμε στην τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 μαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 Τζιν Λάμπερτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23, δύο τμήματα. Α, συγγνώμη, ένα τμήμα, λέει η Πρόεδρος. Ένα τμήμα. Από το encourages μέχρι το gas extraction activities, το δεύτερο τμήμα είναι μη παραδεκτό. Υπέρ λοιπόν του πρώτου τμήματος τροπολογίας 23, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 7, συμβιβαστική F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 μπουλόν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 29 της συγχύτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 διουλών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 μπουλό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης Ποιος δεν έχει κάρτα. Έχουν όλοι κάρτα. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία, η ηλεκτρονική. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 8 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ωραία. Λοιπόν, όπως σας είχα πει στην αρχή της ημερήσης διάταξής μας, θα ψηφίσουμε τώρα τα, ε, το σχέδιο επιστολής ε, ε, για την κινητοποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών, η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει ήδη αποφασίσει για την κινητοποίηση του συγκεκριμένου Ταμείου Προσαρμογής ε, στην ε, ε, παγκοσμιοποίηση. Σας προτείνω λοιπόν, για να διατηρηθεί καλή τάξη των πραγμάτων, να ψηφίσετε κι εσείς τα συγκεκριμένα... τις συγκεκριμένες επιστολές. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση Πρόκειται για το σημείο 17 της κινητοποίησης ε, του Ταμείου για την προσαρμογή στην, στην παγκοσμιοποίηση, συγγνώμη, ε, για, ένα, ε, για ένα ναυπηγείο. Συμφωνείτε? Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομοφόνος. Η επιστολή. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση που αφορά την χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης για την η περίπτωση Glass Fiber από τη Δανία. Έγινε μια προφορική τροποποίηση τελευταία στιγμή για να λάβουμε υπόψη μας την πραγματικότητα, τον τρόπο λειτουργίας δηλαδή αυτή της βιομηχανίας που χρησιμοποιεί η ολική ενέργεια, την ολική ενέργεια που μας αφήνει λίγο έτσι άναυδους. Έχω προτείνει μια πρώτη προφορική τροπολογία ε, διότι κάναμε και κάποια συνεργασία με τις πολιτικές ομάδες και ζητούμε ε, να γίνει μια αλλαγή του κειμένου. Θέλετε να σας διαβάσω την αλλαγή. Ωραία. Τονίζει ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό είναι μια προσθήκη που ζήτησαν οι φιλελεύθεροι. Η παράδοξη κατάσταση όπου οι δεσμεύσει των κρατών μελών για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών δεν αποφέρουν στις εταιρείε ε, τον ίδιο τρόπο όπως ε, για τους ε, ανταγωνιστές τους. Αυτό σημαίνει ότι οφείλεται μάλλον στο γεγονό ότι δεν έχουν ενταχθεί πλήρω στην βιομηχανική στρατηγική τη Ένωση. Δεν υπάρχουν ε, ε, αντιρρήσει, άρα ψηφίζουμε υπέρ. Κατά, από, ε, υπέρ κατά αποχές μετά εγκρίνεται. Έχουμε μια άλλη προφορική τροπολογία που προτείνουν οι πράσινοι. Σας την έχουμε μοιράσει και αυτή. Θέλετε να την ξαναδιαβάσω. Θα την ξαναδιαβάσω τονίζει ότι η ολική ενέργεια είναι ουσιαστική για να πετύχουμε τους στόχους ε, του 2020 όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια. Επίσης εκφράζει τις ανησυχίες τους ότι το ε, ταμείο, τη χρηματοδότηση μάλλον από το ταμείο ε, χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων που εργαζόντουσαν στο παρελθόν σε, στις πράσινες βιομηχανίες έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν σε άλλους τομείς και ζητά από την Κομισιόν τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να αναπτυχθούν πράσινες θέσεις απασχόλησης ε, ευθυγραμμιζόμενοι με τη στρατηγική του 2020. Εφόσον υπάρχουν αντιρρήσει όμω, δεν μπορούμε να αντιψηφίσουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Επομένω, ψηφίζω, ε, προτείνω να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο με την τροπολογία που σα διάβασα στην αρχή, υπέρ κατά αποχέσα Αυτή η δεύτερη επιστολή εγκρίνεται. Τώρα, Πάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, εφόσον ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες μας για σήμερα. Στο σημείο, της, ε, στο σημείο 9 δίνω το λόγο στον κύριο Dirk Sterks για να εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες στην γνωμοδότησή του που αφορά την ε, γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ίντα και έχει σαν θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Μια εμπορική ανισορροπία. Ευχαριστώ τους συναδέλφους καταρχάς για την εξαιρετική συνεργασία. Ε, κάναμε μια συνεργασία όλοι μας για να συζητήσουμε για τη συμβιβαστική πρόταση. Ε, βέβαια για την παράγραφο 5 δεν έχουμε κάποια συμβαστική τροπολογία. Λοιπόν, να στα διακόψω για λίγο έτσι ώστε όσοι να, να φύγουν να φύγουν για να μπορούμε και να συζητήσουμε με ηρεμία. Πρόεδρε, θα σας πρότεινα και εγώ το ίδιο λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, οι συνάδελφοι που θέλουν να φύγουν και κακώς κάνουν που θέλουν να φύγουν, αλλά τουλάχιστον να το κάνουν σιωπηλά. Όχι, τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, μπορώ να συνεχίσω. Υπάρχει μία συμβαστική τροπολογία για την παράγραφο 5. τι γίνεται για τις επενδύσεις της δικές μας στην Κίνα και για τις επενδύσεις των Κινέζων εδώ. Για, εδώ, για, σε αυτή, για την ε, συμβαστική τροπολογία δεν υπήρξε συμφωνία. Όμως ε, για, τις για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει πρόβλημα. Για τη δεύτερη παράγραφο που αφορά το κοινωνικό ε, σύστημα της Κίνας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Γκουτιέρες, τον συνάδελφο Γκουτιέρες, ε, και είναι γιατί είναι ευελιξία τους, διότι ε, η τροπολογία που προτείνουν ε, λαμβάνει υπόψη το υπάρχον κείμενο. Για την παράγραφο 3 που αφορά την ευθύνη της Κίνας σαν μια παγκόσμια οικονομία, σαν μια, παγκόσμια, σαν μια μεγάλη χώρα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα αυτό όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη και τον, ε, την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τους όρους εργασίας και την τήρηση των κανόνων του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Ε, ε, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι Κουτιέρες, Μαν και Λίνε. Νομίζω ότι τελικά καταλήξαμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο εμπλουτίσαμε και με τις προτάσεις των συναδέλφων. Τώρα, για τη νέα παράγραφο. Εδώ προσπαθήσαμε όχι για την τροπολογία γάμα καλύτερα. Να σας πω ότι Υπάρχουν ε, κάποιες τροπολογίες ε, τις οποίες προσπάθησα να λάβω υπόψη μου. Αλλά είναι δύσκολο το έργο γιατί υπήρχαν διστάμενες απόψεις. Τέλος πάντων, ελπίζω να συμφωνούν όλοι με το κείμενο το οποίο παρουσίασα ε, για την τροπολογία 60 τώρα του κυρίου Μέρφυ Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Κίνα είναι κάπως αυστηρή όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπάρχουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνδικαλιστές. Ε, εγώ το είχα εκφράσει με πιο γενικό τρόπο αυτό. Ο κύριος Μέρφυ όμως δεν συμφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη με την τροπολογία 60 στη συμβιβαστική τροπολογία. Άρα η τροπολογία 60 θα ψηφιστεί ξεχωριστά. Συμφωνώ με το περιεχόμενο μεν της τροπολογίας, αλλά θεωρώ ότι είναι κάπως περιοριστικό. Εάν μιλάμε μόνο για τα δικαιώματα των συνδικαλιστών. Εμείς πιστεύουμε ότι η νομοθεσία της Κίνας τον τελευταίο καιρό είναι πολύ πιο, έχει γίνει πολύ πιο αυστηρή, έχει γίνει πολύ σκληρή και όπως είπε και ο κύριος Μέρφυ έχουν περιοριστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα στην Κίνα. Ε, τέλος αυτά για την συμβαστική τροπολογία γάμα Επίσης, για τον κοινωνικό διάλογο ανάμεσα στην Κίνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε ότι μέσα στα πλαίσια αυτού του διαλόγου υπάρχουν κάποια κοινωνικά στοιχεία, κάποια κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν ε, κοινωνικά δικαιώματα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και να μιλήσουμε και για συνθήκες εργασίες, για εργατικά αντικείμενα, για ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών. έτσι ώστε, το διεθνε... έτσι ώστε να γίνονται ε, σεβαστοί οι κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Τέλος πάντων, προσπάθησα να συνοψίσω και να λάβω υπόψη μου όλες τις ε, προτάσεις που ακούστηκαν και ελπίζω ότι οι συμβαστικές τροπολογίες θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε την ε, μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Πάντως πιστεύω ότι δεν πρέπει να βαρύνουμε ιδιαίτερα την γνωμοδότησή μας, διότι ε, υπάρχουν 60 τροπολογίες οι οποίες ε, έχουν υποβληθεί. Αν τις προσθέτουμε όλες αυτές στο κείμενο, σίγουρα θα υπάρχουν επακαλύψεις και θα έχουμε μια γνωμοδότηση ε, η οποία θα είναι κάπως βεβαρημένη θα έλεγα. Και δεν θα έχουμε έτσι μια σφαιρική εικόνα. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν στο κείμενο και ποια όχι. Ελπίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση σαφή και εύχριστη. Ευχαριστώ τον εισηγητή, λέει η πρόεδρος, ο κύριος Αλμέρ. Ευχαριστώ και επιτρέψτε μου παραδοσιακά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη σκληρή δουλειά του και την ιδιαίτερα φιλική αντιμετώπιση των συμβαστικών τροπολογιών. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς η ομάδα μου δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξει είτε τις συμβαστικές τροπολογίες είτε την έκθεση ως σύνολο. Είναι μια ξεπερίεργη περίπτωση επειδή πολλά από αυτά που λέει η έκθεση είναι απόλυτα ομαλά, κανονικά και λογικά και θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά. Η αντίρρησή μας είναι όχι επειδή είναι στραβά αυτά ή είναι λάθος και δεν τα δεχόμαστε, αλλά εξετάσει θέματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου που εκπροσωπούμε και της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Και το να ε, δείχνουμε τους Κινέζους με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά κάτι το υβριστικό και το ιταμό. Βρισκόμαστε εδώ και προειδοποιούμε σε σχέση με το χάσμα μεταξύ πλουσίων και πτωχών ε, τους ε, Κινέζους. Πώς θα αισθανόμαστε αν γινόταν το αντίστροφο, αν γινόταν παράπονο και φραζόταν παράπονο για το χάσμα των πλουσίων και των φτωχών. Ασκούμε επικρίσεις στους, ε, στους Κινέζους επειδή λέμε η φτώχεια και πληθωρισμός και τα λοιπά δημιουργούν προβλήματα. Τα λέμε όλα αυτά όταν βρίσκονται διαδηλωτές στους δρόμους της Αθήνας για τα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί στον ελληνικό πληθυσμό. Είναι αξιοπερίεργο το ότι φερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα αναμέναμε οι Κινέζοι να επικρίνουν τους δικούς μας τρόπους εμείς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Εντάξει, να ασκηθούν επικρίσεις στους Κινέζους εκεί όπου πρέπει να ασκηθούν τέτοιες επικρίσεις σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Κίνα. Αλλά να δακτυλοδείχνουμε τους Κινέζους και να κάνουμε κατηχήσεις και μαθήματα όταν έχουμε προβλήματα εμείς, ε, είναι κάτι το πραγματικά που δεν οδηγεί πουθενά, είναι αντιπαραγωγικό. Η ομάδα μου λοιπόν θα καταψηφίσει αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Τόμας Μαν, μετά ο κύριος Θέρκας. Ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Ναι, το ότι ε, πήρε χρόνο, ναι, αλλά παίρνουμε και προτάσεις ε, από τους συναδέλφους που θεωρούμε ότι είναι θετικές και βρισκόμαστε σε κάτι το οποίο μπορούμε να επισκοπήσουμε και να εργαστούμε θετικά. Είναι σημαντικό να μπορούν να υπάρχουν και συμβιβασμοί. Κάποιοι είπαν ότι, κάποιος είπε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι για αυτά τα θέματα εμείς, θα έπρεπε ίσως για δικαιώματα των ανθρώπων να πούμε έχουμε και τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Ο Ρότζερ είπε δεν μπορεί να προτείνουμε παντός του επιστητού προτάσεις. Αν δούμε την τροπολογία 16 που λέμε η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας έχει ξεχωριστές διατάξεις και κανόνες και που ε, θεσπίζει. Συγγνώμη, είναι μια μεγάλη και ισχυρή χώρα η Κίνα. Ωστόσο όμως είναι μέλος του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Μέλος ε, ενός παγκόσμιου οργανισμού πρέπει να τηρεί τους κανόνες και κανονισμούς αυτούς και πρέπει να συμμορφώνεται με αυτούς. Λοιπόν, σε σχέση με μια χώρα που δεν έχει συνηθίσει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται προς άλλους, νομίζω από κοινού έχουμε βρει μια καλή πορεία. Χωρίς να είμαστε ξερόλες και να κάνουμε κατηχήσεις, αλλά να είναι σεβαστοί οι κανόνες. Να μην υπάρχουν ε, προβλήματα σε σχέση με τις μειοψηφίες, ε, να υπάρχουν κοινέ κοινές ε, που θα γίνονται σεβαστές και είμαι ικανοποιημένος για αυτό το οποίο έχουμε ως αποτέλεσμα από την εργασία του Dirk Sterks και δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι εκτός ε, ε, πραγματικότητας. Συγκεκριμένες προτάσεις ε, διατυπώνονται και συγχαρητήρια θα ήθελα να πω και κάθε επιτυχία εύχομαι. Ο κύριος Θέρκας τώρα παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Η σοσιαλιστική ομάδα πρόεδρε ακολουθώντας τις ε, ενδείξεις τη Ρωμανοπλών. Πρέπει να καταδείξει την γενική συμφωνία της ε, και να ευχαριστούμε πολύ για αυτή την έκθεση και την προσπάθεια που έγινε για να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Ε, εμείς υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Όχι επειδή αντανακλώνται όλες τις θέσεις της ομάδας μας, αλλά επειδή με τους συμβιβασμούς το σημαντικό στο σώμα δεν είναι να έχει κανείς δίκιο σε όλα, αλλά να μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο εφικτό όλοι, βελτιώνοντας ένα κείμενο. Αυτό είναι συμβατό και σε κάποια σημεία παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι μπορεί να έχουμε αντίθετη άποψη. Υπάρχουν σημεία όπου σε σχέση με την πρόοδο όσον αφορά την ε, ε, απώλεια θέσεων ε, εργασίας, όσον αφορά τις αναδιόμενες χώρες, δεν έχουμε προτίμηση ούτε για το αρχικό κείμενο ούτε για τις συμβαστικές τροπολογίες. Πρόκειται για πράγματα τα οποία είναι ε, συζητήσιμα, εν πάση περιπτώσει. Η ομάδα μας ε, θέλει να είναι υπεύθυνη στις θέσεις που θα υιοθετεί. Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα σε κάτι το οποίο αναφέρθηκε πιο πριν και που είναι πάντα ευαίσθητο. Δεν υπάρχει όμως καμιά αμφιβολία ότι όταν έχουμε το θέμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα θέματα αρμοδιότητας της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να στρέφουμε το βλέμμα αλλού και να αγνοούμε κάποια πράγματα και να ξεχνάμε ότι οι εταίροι μας σε μια συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να παραβιάζουν οικουμενικές αρχές που ισχύουν στην Ευρώπη και οικουμενικά αποτελούν τμήμα της ε, κοινωνίας των πολιτών και πρέπει να είναι σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Και δεν είναι ότι κάνουμε μαθήματα σε κάποιους, αλλά υπενθυμίζουμε ότι αυτή απλά είναι η βάση της συμβίωσης στην διεθνή κοινότητα και πρέπει να είναι σεβαστά αυτά τα δικαιώματα και οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα και πρέπει να είναι σεβαστά. Υπάρχουν θεμελιώδεις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας για την εργασία των παιδιών για παράδειγμα, για κοινωνικά δικαιώματα που πρέπει να είναι σεβαστές αυτές οι αρχές από όλες τις χώρες χωρίς καμιά εξαίρεση. Η σοσιαλιστική ομάδα δεν θέλει να πάει πιο πέρα από αυτά, αλλά αν πρόκειται για μια μεγάλη χώρα πρέπει να είμαστε εξίσου αυστηροί όπως και με μικρές ε, χώρες. Δεν παίζει ρόλο το, μεγα... ή το μέγεθος ε, μιας χώρας σε σχέση με αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να, κοιτάξουμε, να στρέψουμε το βλέμμα αλλού. Δεν είναι το θέμα μόνο να υλοποιούν εκείνοι τις ε, προδιαγραφές και εμείς πρέπει να τις υλοποιούμε. Ακούγονται στο σώμα κάποιες φωνές και παρατηρήσεις που είναι κατά του να υπάρχουν παρατηρήσεις επί άλλων για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Δεν είναι για την υλοποίηση εκτός Ευρώπης των κανονισμών και των διατάξεων αλλά και στην ίδια την Ευρώπη να υλοποιούνται οι διατάξεις των Ηνωμένων Εθνών. Καμιά φορά ενοχλεί αυτό το ότι δηλαδή για την εφαρμογή του στην Ευρώπη δημιουργείται θέμα. Η ομάδα μας λοιπόν επιμένει σε αυτή την πτυχή επίσης. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει. Όμως, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επιστρέψω σε κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι ένα σημείο πάρα πολύ ευαίσθητο και το οποίο δεν διαλευκάναμε στη συζήτηση που είχαμε και ούτε θα το λύσουμε και στην ψηφοφορία αύριο. Οι συμβαστικές τροπολογίες όταν καταλήξουν κάπου πρέπει να γίνονται σεβαστές διότι αντιπροσωπεύουν τις, τους συμβιβασμούς όλων. Όμως γίνεται μια επικίνδυνη υποβάθμιση των εργασιών μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων και σε επίπεδο πολιτών αλλά και σε επίπεδο ανθρώπων αυτών καθεαυτών διότι η Κίνα δεν είναι μια δημοκρατική χώρα δεν γίνονται σεβαστά τα όδη δικαιώματα είτε είναι εργαζόμενοι είτε οι άνθρωποι αυτοί είτε είναι απλοί πολίτες όταν συζητάμε για τα διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν καθημερινά, αυτή είναι μια πτυχή την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η αρμοδιότητα μιας επιτροπής ε, μπορεί να συζητηθεί ε, όταν μιλάμε για την ηθαγένεια, ας πούμε, για το χαρακτήρα του πολίτη. Όμως, είναι και θέματα εργασίας. Και στην φιλελεύθερη κουλτούρα, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και ελευθεριών, στην οικονομική ζώνη και στην εργασία έχει ένα ρόλο και ένα βάρος. Όταν δεν γίνονται σεβαστά αυτά τα δικαιώματα, δεν έχουμε συνέπειες μόνο στις ε, συνθήκες διαβίωσης των ατόμων, ε, των οποίων τα δικαιώματα έχουν αφαιρεθεί, εισάγονται και ε, συνθήκες αθέμη του ανταγωνισμού ανάμεσα στις διάφορες επιχειρήσεις, διότι Προφανώ, οι, οι, οι επιχειρήσεις οι οποίες σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τις από τις άλλες που δεν έχουν κανένα, ε, καμία πρόθεση να σεβαστούν τα δικαιώματα αυτά. Άρα, αυτό δεν λέω ότι έχει να κάνει με την ε, παρούσα συμφωνία, αλλά και για το μέλλον, διότι αλλιώς ε, οι εμπορικές συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες μπορεί να αποτελέσουν ένα εργαλείο για την νομιμοποίηση κάποιων αθέμητων διατάξεων κάποιων διατάξεων που οδηγούν σε αθέμητο ανταγωνισμό. Ήθελα να πω ότι και κουλτούρες που είναι πολύ μακρινές από τη δική μας δεν μπορούν να αγνοούν ότι εάν δεν τηρούνται οι θεμελιώδη, τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν θίγονται μόνο τα άτομα των οποίων ε, θίγονται τα δικαιώματα αλλά και γενικότερα η οικονομική ζωή. Ε, πολύ σύντομα συγχαρητήρια στον εισηγητή για την μεγάλη δεξιοτεχνία κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Οι συμβιβαστικές ε, είναι πολύ καλές, περιλαμβάνουν πολλά, ιδιαίτερα η ΣΥ που αφορά το θέμα κλειδί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αναγκαστική εργασία, ε, πρότυπα περιβαλλοντικά και πρότυπα υγείας και για το μεγάλο θέμα, δηλαδή θα κάνουμε διδαχή στους Κινέζους, όχι βέβαια, αλλά γιατί να μην δώσουμε κάποιες συμβουλές που, ε, να τους μιλήσουμε για διδάγματα από το πικρό μας παρελθόν. Ναι, και μην ανησυχείτε, οι Κινέζοι ε, ακούνε ιδιαίτερα όταν κάνουν τους κουφούς. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Αν όχι, ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Στέρκ ε, για να συνοψίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέλτεμερ ήταν ο πρώτος που πήρε το λόγο. Έφυγε δυστυχώς τώρα. Φαντάζομαι ότι είχε πιο σημαντική συνάντηση να πάει από αυτή. Δεν είναι ότι δεν λένε τίποτα ποτέ οι Κινέζοι. Ότι δεν μας λένε τίποτε. Εγώ ήμουν μέλος για πολύ καιρό της αντιπροσωπείας ε, με την Κίνα και οι Κινέζοι. Πολύ συχνά μας έλεγαν όταν τους ε, προσεγγίζαμε για διάφορα θέματα που υπάρχουν εδώ στο κείμενο, ότι χρειάστηκε να πάρουν αυστηρά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι εμείς πήραμε αυστηρά μέτρα για αυξημένη μεγέθυνση στην Ευρώπη διότι είχαμε πρόβλημα με την ε, μεγέθυνση ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτό μας έλεγαν. Και δεν τα καταφέραμε πολύ με την ολοκλήρωση και την ενιαία αγορά και ήταν πολύ δύσκολο στα πλαίσια του εμπορίου και των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Δεν είναι ότι δεν μας λένε τίποτε οι Κινέζοι. Βεβαίως και τονίζουν τις δυσκολίες που βλέπουν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε στρατηγικοί τους εταίροι τώρα πια. Θέλουμε να συνεχίσουμε και θέλουμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις ε, μαζί τους ε, τώρα για το κοινωνικό πολιτικό σύστημα. Σωστά είναι αυτά που είπαμε. Τώρα πρέπει να δούμε τώρα εδώ ένα μειονέκτημα που βγαίνει σε καλό για την Κίνα. Ε, όλα πρέπει να τα συζητήσουμε μπορούμε να μιλήσουμε για ολοκλήρωση, αλλά αυτή συνεπάγεται κάποιες υποχρεώσεις στα πλαίσια της διεθνούς οικονομίας. Θα τους πούμε τις υποχρεώσεις, θα τους τονίσουμε πού θεωρούμε εμείς ότι ε, ανταποκρίθηκαν και πού όχι. Η Διεθνής Επιτροπή Εμπορίου νομίζω ότι έχει ε, κάποια ευθύνη εδώ. Νομίζω ότι είναι πιο αρμόδια και από εμά ακόμη αν η Κίνα έχει μία θέση που τους διασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αθέμητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ε, δεν είναι πολλά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έχουν ε, μπορικές διάβλους δραστήριες και ενεργές, ενεργούς με την ε, Κίνα και όταν ε, βεβαίως γίνονται επενδύσεις θέλουν κάποια θετική απόδοση των επενδύσεων. Υπάρχουν πολλές εταιρείε και στη δική μου εκλογική περιφέρεια υπάρχουν αρκετές που που μου λένε και θα το συζητήσουμε όταν ε, φτάσουμε εκεί. Υπάρχουν εταιρείε λοιπόν που μου λένε ότι οι επενδύσεις μας εδώ είναι δραστήριες ε, διότι έχουμε εμπόριο και επενδύσεις στην Κίνα και στην Τουρκία και τη Βραζιλία επίσης, όχι μόνο την Κίνα. Υπάρχει λοιπόν κάποια σχέση, ένας σύνδεσμος μια σχέση μεταξύ οικονομικής υγείας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη που εμπορεύονται και επενδύουν όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Κίνα επίσης, για παράδειγμα. Μιλήσαμε για την κοινωνική πολιτική, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το άνοιγμα των συνόρων κλπ. Αυτά τα στοιχεία είναι επίσης σημαντικά, συμφωνώ. Εγώ προσπάθησα να περιοριστώ στα στοιχεία εκείνα τα οποία ε, είναι της αρμοδιότητας της Επιτροπής μας, αλλά ε, νομίζω ότι ο τόνος και η ουσία των τροπολογιών καλύπτουν τα στοιχεία που αφορούν την αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, απασχόληση κλπ. Όλα αυτά τα στοιχεία όμως έχουν άμεση σχέση με τι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνας και δεν πρέπει όλα αυτά να τα βλέπουμε με μάτι αρνητικό. Δεν συμφωνώ με εκείνου που λένε ότι η, ε, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τα προσέξαμε όσο έπρεπε. Δεν συμφωνώ. Μπήκαμε σε πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα στις συμβαστικές τροπολογίες. Ελπίζω αύριο που θα ψηφίσουμε το, την πρόταση ψηφίσματος, η γνωμοδότηση να ε, αντιπροσωπεύει την ε, πλειοψηφία στην Επιτροπή μας. Αυτό θα είναι χρήσιμο και στην τελική έκθεση που θα υποβάλει ο συνάδελφος για το Διεθνές Εμπόριο. Ευχαριστούμε κυρία Σιγητά. Η συζήτηση αυτή ακολουθεί αυτό που αποφασίσαμε για το, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι περίπου η ίδια συζήτηση, γιατί στο πλαίσιο αυτού του εργοστασίου παραγωγής αιωλικής ενέργειας, ε, στη Δανία μιλάμε για μια ενέργεια η οποία είναι πολύ σημαντική για το μέλλον. Το επιχείρημα για το κλείσιμο είναι περισσότερες επενδύσεις στην Κίνα για να είναι πιο κοντά στην κινέζικη αγορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για το οποίο δεν πρέπει να είμαστε αφελείς ως Ευρωπαίοι. Αύριο θα ψηφιστεί η γνωμοδότησή σας, όπως είπατε και εσείς ο ίδιος. Ήθελα απλώς να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι Κρίθηκαν μη παραθεκτές κάποιες τροπολογίες γιατί δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της δική μα Επιτροπής αλλά τη Επιτροπή Νομικών Υποθεσέων διεθνού Εμπορίου ε, πολιτισμού και περιβάλλοντος και επειδή μας απασχολεί, μας απασχολεί πολύ να μην μπαίνουν στα χωράφια μας οι άλλες επιτροπές βλέπετε ότι θα είμαι πολύ αυστηρή να ευζηφίσουμε πράγματα τα οποία δεν καλύπτονται από τις αρμοδιότητές μας και σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν ε, για την κατανόησή σας, ε, για το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές 10 τροπολογίες. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και... Θα το ψηφίσουμε κιόλας αύριο θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον εισηγητή γιατί δεν θα μπορώ να είμαι εδώ. Αλλά δεν πειράζει, θα είναι εδώ η αντιπρόεδρος, οπότε όλα θα πάνε καλά. Και πάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, που είναι μια ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο της έκθεσης ε, της ε, συναδέλφου μας ε, Ρεζίνα Μπάστος, για μία από τις βασικές πρωτοβουλίες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Πρόκειται για την ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Πριν δώσω το λόγο στους πέντε προσκεκλημένους μας, ε, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία τους, θα ήθελα να δώσω για λίγο το λόγο στην εισηγήτριά μας για να μας αναφερθεί στο γενικό πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Έχετε το λόγο κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινώ ευχαριστώντας, ευχαριστώντας για την αποδοχή της πρόσκλησης από πλευράς των αγορητών για αυτή τη δημόσια ακρόαση για την ατζέντα για τις νέες δυνατότητες και την απασχόληση, ε, νέες δεξιότητες και απασχόληση. Είμαι πισμένη ότι οι παρουσιάσεις που θα ακούσουμε από τους αγορητές θα είναι αξιόλογες παρουσιάσεις για να εμβαθύνουμε και να γνωρίσουμε τις διαφορετικές απόψεις ως προσεγγίσεις στο πανόραμα της σκηνής των εργασιακών θεμάτων για την Ευρώπη για τα επόμενα δέκα χρόνια. Στην έκθεση που το σχέδιο έκθεσης σας είναι γνωστό, έχουμε ως κυριότερους στόχους να δώσουμε απαντήσεις ακριβώς στις προκλήσεις της απασχόλησης και τις δεξιότητες και προσόντα που απαιτούνται για αυτή την απασχόληση, διαμόρφωση του πλαισίου απασχόλησης. Και θέλουμε να ανταποκριθούμε στην φιλοδοξία της στρατηγικής 2020 για την Ευρώπη, να πετύχουμε το 75% απασχόλησης ανδρών και γυναικών ε, στο ηλικιακό ε, φάσμα, φάσμα 20 έως 60 ετών. Έχουμε προκλήσεις που πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε αυτές. Προκλήσεις ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, επιτυχή πολιτική απασχόληση σε σχέση με την ανακοίνωση κιόλας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά, αλλά και μια προσέγγιση στην έκθεσή μου ξεχωριστή υπό του να υπογραμμίζουμε την ε, ε, αντίθεση, ας το πω έτσι, την διαφοροποίηση σε σχέση με οικουμενικές ή παγκοσμιοποιημένες ε, λύσεις. Κάθε χώρα έχει τις ειδικές της ιδιομορφίες και πρέπει ανάλογα με αυτές τις δικές της ιδιομορφίες και ανάγκες να σχεδιάζονται οι απαντήσεις. Και έτσι πρέπει να δούμε και να δράσουμε για τα επόμενα χρόνια. Επίσης να δώσουμε απάντηση για την προαγωγή, την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ανοίγοντας ε, δυνατότητες, δημιουργώντας ε, μια γέφυρα ώστε να γεφυροποιήσουμε την ζήτηση και την προσφορά σε σχέση με την αγορά εργασίας, βλέποντας τις ανάγκες σε σχέση με την κατάρτιση και την εκπαίδευση και την παιδεία, τις ανάγκες που έχει ο χώρος της ε, ε, εργασίας και οι επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και την αναβαθμισμένη ποιότητα στις θέσεις απασχόλησης, στην εργασία. Κύριοι παράγοντες της έκθεσής μου, δεν θέλω να μακρηγορήσω υπερβολικά, επαρκούμε σε αυτές τις γενικές γραμμές διαρθρωτικά της έκθεσης ε, που έχω πρόθεση να συνεχίσω να βελτιώνω και να διαρθρώνω με την συνεισφορά των επαϊόντων που θα ακούσουμε και με τις τροπολογίες των συναδέλφων. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους αγορητέ που προσκαλέσαμε στην ακρόασή μας και προσβλέπω ιδιαίτερα στο να ακούσω τα μηνύματα και τις ιδέες που έχουν να μα δώσουν για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο η Θα ήθελα να απλώς να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στους ε, προσκεκλισμένους μας με, τον, με τη σειρά που μου πρότειναν. Επομένως, ε, την τιμή και το προνόμιο να ξεκινήσει ε, έχει η Business Europe που σήμερα την εκπροσωπεί η κυρία Έλενα Στρίγκραντ που είναι σύμβουλος για τις κοινωνικές υποθέσεις. Πέντε με 7 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι προνόμιο αυτό. Καταρχήν να πω ότι στα διάφορα θέματα που προτάθηκε να συζητήσουμε υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα που μας απασχολεί πολύ γιατί είναι αυτό που θεωρούμε το πιο σημαντικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την επίτευξη του στόχου απασχόληση 75%. Δηλαδή η ευελιξία με ασφάλεια, η εγκυρότητα της αρχής αυτής, εποχή κρίσης. Ε, είναι σαφές ότι η ευελιξία με ασφάλεια έπαιξε κέριο ρόλο στην κρίση. Βλέπουμε ότι χώρες που ήδη έχουν εφαρμόσει τις αρχές εδώ είναι εκείνες που βγήκαν λιγότερο ταλαιπωρημένες από την κρίση, όπως η Ολλανδία. Ε, πολλοί θα πούν ότι τη σήμερα ημέρα αυτό που λένε οι εργοδότες είναι ευελιξία, ευελιξία, ελαστικότητα. Η ευελιξία με ασφάλεια είναι ένα πακέτο. Υπάρχει το κομμάτι της ασφάλειας και της ευελιξίας. Είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Υπάρχει ανάγκη αύξηση της ευελιξίας, αυτό το πολεμούν πολύ και μας εκπλήσει. Γι' αυτό θα ακούσετε εργοδότες να υπενθυμίζουν, να τον επαναλαμβάνουν τη σημασία του θέματος αυτού. Δεν θα με εξαίρεση εγώ, αρχίζω λέγοντας ότι αν δεν υπήρχε η εσωτερική ευελιξία τώρα με την ε, πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ευελιξία με την έννοια των βραχυπρόθεσμων μορφών απασχόλησης, τότε θα είχαν χαθεί και άλλα μερικά εκατομμύρια θέσεων εργασίας. Είναι γεγονός. Ξέρουμε ότι στη Γερμανία το 2009, σύμφωνα με το Ινστιτούτο τη αγορά εργασία, 1,2 εκατομμύρια θέσεων εργασία διεσώθησαν λόγω αυτών των καινούριων μορφών εργασία. Και αν δούμε, ας πούμε, και την εξωτερική ευελιξία, είναι και αυτή εξίσου σημαντική, γιατί οι εταιρείε ζουν σε μια πραγματικότητα αστάθειας και αβεβαιότητας. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα για να μην έχουμε ανάπτυξη χωρίς θέσεις εργασίας είναι να αρχίσουν οι προσλήψεις πάλι για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια τα σχετικά και οπωσδήποτε θα πρέπει να δώσουμε όλες τις λύσεις. Δεν, δεν, μπορούμε να έχουμε πια ε, αόριστου χρόνου συμβάσεις, γιατί δεν υπάρχει η ε, ανάπτυξη ακόμα που τόσο χρειαζόμαστε. Ένα στοιχείο της ε, ευελιξίας με την ασφάλεια που κατέδειξε την ε, σημασία του είναι η διαβίου μάθησης δηλαδή η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Και είναι ενδιαφέρον που βλέπουμε ότι ένας λόγος γιατί η Ευρωπαίοι εργαζόμενοι απολύονται λιγότερο από τους Αμερικανούς είναι ότι οι εργοδότες επένδυσαν στις, στις ε, δεξιότητές τους. Έχουν πια δεξιότητες πολύτιμες για τους εργοδότες και θέλουν να τους κρατήσουν γι' αυτό όσο μπορούν. Και αν υπάρχει κάτι που πρέπει και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας να μην μειώσουν είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση, γιατί αυτό είναι μια ζωτική επένδυση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα τελευταία είδαμε αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβάνοντας την κατάρτιση που γίνεται και ενδοεπιχειρησιακά. Ανέφερα δύο πυλώνε τη ευελιξία με την ασφάλεια. Όπως ξέρετε όμω, αυτό είναι συμφωνία πακέτο και σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουμε σε ενεργές πολιτικές τη αγορά εργασία αναδιάρθρωση συστημάτων κοινωνικών επιδομάτων για να λειτουργούν και να είναι και βιώσιμα. Γιατί όταν μιλάμε για την ασφάλεια θα πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να είναι βιώσιμη, θέλουμε βιώσιμη ε, ασφάλεια, όχι μόνο μέσο αλλά και, ε, και μακροπρόθεσμα για τις επόμενες γενναίες. Και για να το πω έτσι λίγο ομά, ε, αντιμετωπίζω μια τεράστια μεταρρυθμιστική πρόκληση. Τώρα πάμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας με συστήματα ευελιξίας ασφάλειας και δεν έχουμε χρόνο για να τα κάνουμε όλα αυτά. θα ήθελα να να παραπέμψω σε μια μεγάλη ανάλυση που έκανε το Business Europe, προσπάθησε δηλαδή να κάνει διάγνωση της κατάστασης ε, της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Και φαίνεται ότι για παράδειγμα οι δυσκολίες των κρατών μελών κατά την κρίση αυτά δεν είναι προσωρινά πράγματα. Έχουμε δομικές, ε, δομικά προβλήματα, έχουμε αντιστοιχεία μεταξύ ε, προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Έχουμε ε, χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας που ε, λάμβανε χώρα επί σειρά ετών. Αυτά είναι συμπτώματα υποκείμενης δομικής αδυναμίας. Θα πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά. Και τώρα είναι η ώρα της αλήθειας. Στα κράτη-μέλη πρέπει να τα ρυθμίσεις. τα εθνικά μας τα προγράμματα δεν ε, αντικατοπτρίζουν, δεν δείχνουν ε, τόσο μεγάλες ε, μεταρρυθμίσεις όσο χρειάζονται. Αυτό είναι μεγάλο μέλημα και ανησυχία για μας. Γιατί εκατομμύρια Ευρωπαίοι παραμένουν άνεργοι, για να μην μιλήσω και για το οξύτατο πρόβλημα των νέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε σε προσώπους των συνδικάτων και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Λούκα Βισεντίνη, ο γραμματέας της Νομοσπονδίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, ε, την πρόσκληση που μας στείλετε για να συμμετέχουμε σε αυτή την ακρόαση. θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα την ε, συνεισφορά μας. Όταν το 2008 ξεκίνησε αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, ένα agenda for new skills and jobs ε, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 η οικονομική κρίση μόλις είχε ξεκινήσει. Αυτή η πρωτοβουλία πρότεινε φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την ανάπτυξη της ε, απασχόλησης ε, των ποσοστών παιδείας, καταρχικής κατά, κατάρτισης, διαβίου κατάρτισης, μείωση των, της εγκατάλειψης του σχολείου. Βέβαια μετά την κρίση όλοι, αυτοί οι δείκτες επιβαρύνθηκαν. Η ανεργία στην Ευρώπη αυξήθηκε, οι κατηγορίες οι οποίες επλήγησαν περισσότερο ήταν οι νέοι, οι με μεγαλύτερες εργαζόμενοι, τα άτομα με, το, χαμηλότερη εκπαίδευση και λιγότερα επαγγελματικά προσόντα. Οι αναδιορθώσεις από στις οποίες οδήγησε η κρίση προσθέθηκαν στα προβλήματα που σχετίζονταν με την καινοτομία, με τις κλιματολογικές αλλαγές, με τις διάφορες αναρθριαθρώσεις των τομέων, στην πίεση της του παγκόσμιου ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές. Ε, καθορίστηκε ένα πλήρες, ένα πλαίσιο το οποίο οδήγησε στην επιβάρυνση και στην επιδίνωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων που οφείλονταν στην, στον περιορισμό των πόρων που προσανατολίζονταν στην κατάρτιση για την ένταξη και στην επαγγελματική ενημέρωση. Ε, σε, αντίθεση με τους στόχους που είχαν οριστεί για τη στρατηγική της Ευρώπης του 2020 και στην ατζέντα για τα νέα προσόντα και, για την και εργασία, οι πολιτικές στην στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση ε, ε, υπέστησαν ε, μια επιβράδυνση σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα οι πολιτικές της ε, Flex Security που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε μια αύξηση των θέσεων απασχόλησης ε, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη κινητικότητα και ένα δίκτυο προστασίας, κοινωνικής προστασίας δεν πέτυχαν τους στόχους τους. Μειώθηκαν συνολικά οι θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και αυξήθηκαν οι οι, οι θέσεις ε, απασχόλησης ε, ε, που ήταν περιορισμένης χρονικής διάρκειας, που δεν ήταν καλά και που χρειαζόντουσαν χαμηλότερα προσόντα. Άρα είδαμε ότι στην μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών προφανώς οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν οδήγησαν στα αποτελέσματα τα οποία θα θέλαμε. Άρα θα πρέπει να επανεξετάσουμε όλη την στρατηγική μας. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι και τα εργαλεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα για τα νέα προσόντα και ε, αργασίες θα πρέπει να εστιάσουν καλύτερα την, τη δράση τους ε, και να προσαρμοστούν βέβαια και στην ε, κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία έχει ορίσει κάποιες βασικές προτεραιότητες. Καταρχάς θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια αρχική παιδεία υψηλού επίπεδου και να περιορίσουμε τον αριθμό της εγκατάλειψης, τον αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν το, σχολείο, εγκαταλείπουν το σχολείο. Η αρχική εκπαίδευση είναι σημαντική όχι μόνο για την προσωπική ανάπτυξη, αλλά επίσης γιατί θέτει τις βάσεις για πολίτες οι οποίοι είναι ενεργοί, ε, της βάσεις για μια κοινωνική ένταξη και για την ε, επιτυχία της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ίση προσέγγιση, ισότιμη προσέγγιση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση θα πρέπει η κατάρτιση να είναι ε, προσβάσιμη, προσπελάσιμη και κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να επικυρώσουμε την ε, επίσημη αλλά και την ανεπίσημη κατάρτιση. Ε, αυτό προσφέρει ευκαιρίες ενσωμάτωσης στην κοινωνία εν γέννη και στην αγορά εργασίας συγκεκριμένα. Βοηθάει την πρόληψη της ανεργίας των εργαζομένων που έχουν προσόντα αλλά χωρίς κανένα τίτλο τίτλο Θα πρέπει να διευκολύνουμε το πέρασμα από την αρχική κατάρτιση στο χώρο εργασίας ε, θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμη την, την κατάλληλη χρηματοδότηση είναι αντιπαραγωγικό για τι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να περιορίσουν τους πόρους για την παιδεία και την κατάρτιση, διότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται από, τις, από τα προσόντα των πολιτών, από των, εργαζομένων αλλά και των άνεργων. Οι, οι εργοδότες ψάχνουν ε, πάντα να βρουν εξειδικευμένους εργαζόμενους και θα πρέπει να αναγνωρίσουν και τη δική τους ευθύνη στην υποστήριξη της, ε, της επαγγελματικής κατάρτισης σαν μια επένδυση για την ανάπτυξη ανάπτυξη, συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο ε, για την ε, διαβίου ε, κατάρτιση. Η συμμετοχή των συνδικάτων είναι ένα σημείο κλειδί, ένα στοιχείο κλειδί για την διαχείριση και τον έλεγχο των δημοσίων πολιτικών και των συστημάτων κατάρτισης θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες για την επαγγελματική κατάρτιση ειδικότερα στον χώρο εργασίας, επίσης θα πρέπει να λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πρωτοβουλίες αλλά και τα ευρωπαϊκά εργαλεία που αφορούν την κατάρτιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες συγγνώμη, και ε, πάρα πολλά εργαλεία για να υποστηρίξουν την δραστηριότητα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια της ατζέντα για νέα προσόντα και εργασίες. Για να ολοκληρώσω ωστόσο η συνομοσπονδία μας θεωρεί ότι όλοι αυτοί οι στόχοι ε, αποτελούν ένα ε, απαραίτητο, μια απαραίτητη προϋπόθεση ε, για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να δράσουν όμως όλοι, όλα αυτά τα, όλες τις δυνατότητες και πρωτοβουλίες ε, ε, αυτόνομα. Θα πρέπει να δράσουμε συλλογικά. Αυτό το οποίο, μας, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να δράσουμε συλλογικά, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις θέσεις απασχόλησης, θα πρέπει μέσω της οικονομικής διακυβέρνησης και μέσω του Europlus Pack να ε, προχωρήσουμε. Χρειάζονται διάφορα μέτρα για να, για να σώσουμε τις διάφορες χώρες, για τα Eurobond, για τα ευρωομόλογα παραδείγματο χάρη. Ε, θα πρέπει να ε, σταματήσουμε τις πολιτικές περικοπής των μισθών, ακόμα και τα προγράμματα τα εκπαίδευση και κατάρτιση ε, ε, υφίστανται περικοπές. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Επίση, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τον κοινωνικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους σε συνεργασία με τον τομεακό κοινωνικό διάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, ο Κριστιόν Λετμάιερ. Ε, είστε ο ε, ενεργεία διευθυντής του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Μπερές, ευχαριστώ κυρία Μπάστος, ευχαριστώ πολύ το Κοινοβούλιο για την πρόσκλησή του. Η αναντιστοιχία που αναφέρθηκε προηγουμένως είναι όταν έχουμε υψηλά ποσοστά ανεργίας ή ε, και παράλληλα έχουμε και πολλή διαθεσιμότητα θέσεων απασχόλησης, παράλληλα μερικές φορές το ένα με το άλλο. Ε, Παρ' όλα αυτά σε 27 χώρες μέλη επιχειρήσεις δεν βρίσκουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τις ανάγκες τους. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Η αναντιστοιχία υπάρχει ε, στις θέσεις απασχόλησης όταν τα προσόντα των ε, εργαζομένων είναι πολύ διαφορετικά από τις ανάγκες της ε, ε, θέσης εργασίας. Αυτό περιορίζει πάρα πολύ τις δυνατότητες που έχει ο εργαζόμενος και έχει και ένα αποτέλεσμα βέβαια στην παραγωγικότητα. Η απασχολησιμότητα είναι προϋπόθεση για την ενσωμάτωση στην κοινωνία. Όμως δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση. Τα προσόντα, οι δεξιότητες, οι ικανότητες, υποβαθμίζονται όσο περνάει ο καιρό και πρέπει να ενημερώνονται, να αναπτύσσονται. Υπάρχουν διαρθρωτικέ αλλαγέ, τεχνολογική πρόοδο και αυτό αυξάνει την ανάγκη για ε, συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και διαβίου εκμάθηση. Όλο και περισσότερο τρόπος ζωής ε, χαρακτηρίζεται από μεταβάσεις ε, μεταξύ περιόδων, από, μετάβαση από τη μία περίοδο ε, απασχόλησης σε μία περίοδο ανεργίας για διάφορους λόγους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες δεξιότητες διαχείρισης των σταδιοδρομιών. Ένας από, ένα από τα βασικά στοιχεία αυτής ε, της ε, πρωτοβουλίας είναι ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη αντιστοίχηση των, ε, της προσφοράς και της ζήτησης Χρειαζόμαστε επίσης μια πρόβλεψη των ε, ε, δεξιοτήτων και τα αποτελέσματα πρέπει να ε, είναι εμφανή σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και οι δεξιότητες να είναι διαθέσιμες στους εργαζομένους και τους εργοδότες. Το να υπάρχει μια τέτοιου είδους ευφυΐα στο εργατικό δυναμικό είναι μια προσέγγιση που περνάει από πολλά στάδια περνά μέσα από διάφορε τάσει, τομεακές, επαγγελματικέ, ε, Υπάρχουν επίσης και ιδιαίτερα τάξει, οι οποίε πρέπει να αξιολογηθούν. Ε, υπάρχουν τομεακέ και περιφερειακές ε, εξελίξεις που καταλήγουν στο σχεδιασμό ανθρωπίνου δυναμικού σε μερικές, στις μεμονωμένες οργανώσεις, σε συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να συντονίσουμε τις δομές και είναι προφανές ότι η ενεργό συμμετοχή και η συνεισφορά των εργαζομένων ε, όσων παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση των υπηρεσιών απασχόλησης και των ε, συμβούλων είναι απαραίτητη. Η δική μας δουλειά όσον αφορά την, ε, την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού της αντιστοιχίας είναι μια γενική εικόνα, το να δοθεί μια γενική εικόνα, ένα πανόραμα των δεξιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση του εργατικού δυναμικού. Η ΕΣΚΟ είναι μια προσπάθεια κοινή γλώσσας μεταξύ των ε, ε, μεταξύ της εργασίας και της εκπαίδευσης και ε, αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΚΟ. Έχουμε πολλές, πολλούς εργαζόμενους με, με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και αυτός ε, είναι ο βασικός λόγος ε, της ε, μεγάλης αναλογίας χαμηλής ειδίκευσης εργατικού δυναμικού. Οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι αποσύρονται από την αγορά εργασίας και μερικές φορές ε, οι χαμηλή ειδίκευση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μην ε, ε, ξαναβρίσκουν εργασία αν μείνουν από την αγορά εργασίας εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, επίσης πάρα πολλοί ε, που αφήνουν το σχολείο νωρίς ε, είναι συνήθως άνθρωποι με χαμηλή ειδίκευση που έχουν πολλές, έχουν, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες απασχολησιμότητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό το να φεύγει κανείς από το σχολείο, να καταλείπει καλή στο σχολείο νωρίς, έχουμε διαπιστώσει ως ΣΕΝΤΕΦΟΠ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ήταν άλλωστε κατοικείμενο ακρόαση τον Νοέμβριο του 2010 η βασική μας πολιτική θα πρέπει να είναι να αυξήσουμε τις δεξιότητές τους. Η επαγγελματική κατάρτιση και ε, εκπαίδευση ε, είναι ο σωστός τρόπος ε, για να μπορέσουμε να δώσουμε στην νεολαία που μειονεκτεί ε, κάποια, κάποιες επαγγελματικές προδιαγραφές. Η εκμάθηση δεν είναι μόνο ένας καλός τρόπος ε, για την αύξηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, αλλά εξοικειώνει τους νέους και όλες με τις απαιτήσει του χώρου εργασίας και τους δίνει ικανότητες όπως, για παράδειγμα, ε, ομαδική εργασία, επίλυση προβλημάτων, εστίαση σε συγκεκριμένα καθήκοντα κλπ τους προετοιμάζει για την εργασιακή ζωή. Υπάρχει και μια θεωρητική κατάρτιση με την οποία αν συνδυαστεί δίνει τη δυνατότητα μιας καλής ισορροπίας γνώσης και δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ε, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια επαφής με τους, εργοδότες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης και ε, εκπαίδευσης ε, όλο και περισσότερο συμπεριλαμβάνεται ως είδος ε, εκπαίδευσης και αύξησης των προδιαγραφών που χρειάζεται η αγορά εργασίας γιατί υπάρχει και η δυνατότητα εκμάθησης στο χώρο εργασίας η οποία είναι επίσης πολύ σημαντική παρά το γεγονός ότι μια τέτοιου είδους δυνατότητα συνήθως δίνει ένα χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης. Ε, η ανώτερη εκπαίδευση και η ε, επαγγελματική κατάρτιση δεν αποκλείουν το ένα το άλλο. Ίσως θα έπρεπε να μπορούμε να περνάμε από το ένα στο άλλο μέσω ενός ε, συστήματος, κατάλληλου συστήματος εκπαίδευσης. Πρέπει όμως κάτι τέτοιο να είναι ελκυστικό. Πρέπει να έχουν μια δεξιότητα οι φοιτητές η οποία θα τους χρησιμεύσει κάποια στιγμή στη ζωή τους το να μαθαίνει κανείς το χώρο εργασίας είναι η πιο συχνή και σημαντική ε, μορφή συνεχού συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης ε, και ορίζεται από τις ειδικέ ανάγκες μιας εταιρείας ενός οργανισμού και πρόκειται για ε, αρμοδιότητες οι οποίες δεν είναι πάντοτε επικυρωμένες με κάποιο χαρτί, δεν αναγνωρίζονται και αυτό δεν σημαίνει πολλά για την απασχολησιμότητα του ατόμου αυτού πέρα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει αναγνώριση όλων αυτών των προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο χώρο εργασίας, εκτός δηλαδή του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης, υπάρχει ανάγκη να ε, οικοδομήσει κανείς ολόκληρες σταδιοδρομίες με αυτόν τον τρόπο. με το 2012 τα κράτη-μέλη θα προβούν σε αυτή τη ε, ε, διαδικασία καταχώρησης των πλαισίων εθνικών ε, ε, προδιαγραφών, ε, τα οποία θα συμπεριλάβουν όλα τα είδη των προδιαγραφών, θα αυξήσουν τη διαφάνεια των επαγγελματικών προδιαγραφών στην Ευρώπη και θα δώσουν τη δυνατότητα επικύρωσης των προδιαγραφών αυτών. Θα ήθελα να τονίσω ότι ε, τα νέα ε, ε, εργαλεία που αναπτύσσουμε δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, είναι αλληλοσυμπληρούμενα, ενισχύουν το ένα το άλλο. Να ολοκληρώσω για τη χρηματοδότηση. Ένα σημαντικό, μια σημαντική συνέπεια της ανάπτυξης εφαρμογής των ευρωπαϊκών μέσων και αρχών της επαγγελματικής κατάρτισης ήταν ότι αποτέλεσε ένα μοχλό ε, μεταρρυθμίσεων, ε, τουλάχιστον όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη των ε, συστημάτων επαγγελματική κατάρτισης και κατά τη διάρκεια της κρίσης αυξανόμενα κονδύλια διατέθηκαν, αυξημένα κονδύλια διατέθηκαν σε σχέδια τα οποία βασίζονται σε κοινή χρηματοδότηση. Άλλωστε το ανέφερε και ο συνάδελφος από την ΕΤΟΚ ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα ούτως ή άλλως επηρεάζουν και τη χρηματοδότηση της επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει λοιπόν να βρούμε και νετόμες προσεγγίσεις για να υπάρξει συνεργασία και να λαμβάνονται σωστά υπόψη και τα αποτελέσματα, ε, να υπάρχουν κάποια, κάποιοι τρόποι μέτρησης ε, των αποτελεσμάτων αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ε, εξασφαλίσουμε την ποιότητα της επαγγελματική κατάρτισης και επίσης να υπάρχει και επαρκή ε, επένδυση για την κατάρτιση ε, των ενηλίκων. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μπάρμπαρα Γκέστενμπεργκερ από τη Eurofound. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Μπάσος για την πρόσκληση και την ευκαιρία να σας προσφωνήσουμε σε αυτή την ακρόαση από την Eurofound. Η Eurofound έχει έργο σε αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης. Η flexicurity είναι ένα από αυτά και είναι ενδιαφέρον αυτό. Τονίζουμε το πώς η Business Europe έδωσε έμφαση στην μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πολύ πρόσφατα έχει ερευνηθεί αυτό από το Ίδρυμα και θα βρείτε αναφορά σε σχέση με μια ε, έκθεση για τις επιπτώσεις ε, σε σχέση με αυτή την προσέγγιση. Επίσης, ε, μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την ε, αναφορά της απασχόλησης, ε, αλλά θέλω να αναφερθώ στην στις ίσες ευκαιρίες και τις, τους ίδιους όρους για την απασχόληση που πρέπει να ισχύουν στην ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και ικανότητες για την απασχόληση. Όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα της ποιότητας είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και έχει πολλές ε, συνιστώσεις. Μια καλή θέση απασχόλησης δεν είναι μόνο μια καλοπληρωμένη δουλειά, δεν είναι μόνο μια δουλειά που ε, δίνεται σε χρόνο που είναι βολικός για τον εργαζόμενο έχει ένα πολύ πιο περίπλοκο και σύνθετο χαρακτήρα. Και γι' αυτό η Eurofound ως Ίδρυμα όταν ερευνήσαμε αυτό το ζήτημα βασιστήκαμε και βασιζόμαστε σε ένα πλαίσιο που έχει τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις. Σίγουρα μπορεί να επινοήσει κανείς και διαφορετικά άλλα πλαίσια. Αλλά αυτό το οποίο εμείς δημιουργήσαμε έχει το προτέρημα πρώτα απ' όλα να συζητήσουμε είτε και από τους ερευνητές, αλλά βρέθηκε επίσης και ότι εγκρίνεται από την την τριμερή ε, δομή, δηλαδή τους ε, ε, εντολείς μας, τους εμπλεκόμενους σε αυτό. Πρέπει ως πρώτο σημείο αναφοράς και συμπέρασμα να πούμε ότι είναι το πρώτο στοιχείο τι είναι η μια καλή δουλειά και πράγμα το οποίο είναι μεγάλη πρόκληση ακόμα ως ζήτημα. Ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά η ποιοτική διάσταση έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που αντιμετωπίζουμε και πολλά από αυτά αναφέρονται στο σχέδιο έκθεσης. Για παράδειγμα, η δημογραφική κρίση. Αν θέλουμε να παραμείνουν περισσότερο χρόνο στην απασχόληση οι άνθρωποι, αυτό θα είναι δυνατό να γίνει μόνο αν έχουν ποιοτική ε, ας το πω έτσι συνιστόσα οι θέσεις απασχόλησης και θα είναι ελκυστικές. Αν θέλουμε για τις ε, ευάλωτες ομάδες ε, να λάβουμε υπόψη κάποια πράγματα, κάποια κριτήρια πρέπει να θεσπιστούν που πρέπει να καλύπτονται και αυτό θα πρέπει να μπορεί να αντισταθμίζει την περίοδο εργασίας ε, με εκείνη που ε, ο ε, άνθρωπος δεν θα εργάζεται. Πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη συνιστόσα για την αμοιβή και να ληφθούν υπόψη και οι δεξιότητες και η χρήση των δεξιοτήτων. Η όλη συζήτηση για την flexicurity αφορά επίσης και την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης. Το να έχει κανείς μια θέση με θεμελιώδη δικαιώματα και με την ασφάλιση της ασφάλεια ως προοπτική της απασχόλησής του. Τώρα μια ολόκληρη σειρά πρακτικών θεμάτων. Τι βρήκαμε για αυτές τις συνιστώσεις. Ε, κυρίως θα αναφερθώ στο ερωτηματολόγιο που ε, είχαμε ε, πανευρωπαϊκά. Αυτό που βλέπουμε με τον γυράσκοντα πληθυσμό και την διατήρησή του μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη θέση εργασίας τους το ποσοστό των εργαζόμενων στα 27 κράτη-μέλη που θεωρούν ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τα εργασιακά τους μέχρι τα 60 τους χρόνια αυξήθηκε, έστω και περιθωριακά, από 57 σε 59% μεταξύ του 2000 και του 2010. Ωστόσο όμως από την άλλη πλευρά, ως ήθιστε, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. 70% των εργαζομένων στην Ολλανδία και στη Γερμανία πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους 60. Από την άλλη πλευρά του φάσματος έχουμε τη Σλοβενία με μόνο 26% των εργαζομένων που ρωτήθηκαν πέρσι θα είσαστε σε θέση να εκτελείτε την, ε, τα καθήκοντά σας ε, μέχρι τα 60 σας χρόνια. Μόνο αυτό το μικρό ποσοστό απάντησε ε, καταφατικά και δεν είναι μόνο μια θεωρία, η προσέγγιση, η άποψη αυτό. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει μια πολύ στενή αντιστοιχεία με το πραγματικό ποσοστό των ε, ε, ενεργών εργαζομένων στην ηλικιακή αυτή, ε, ας το πω έτσι, φάση. Τι εξηγεί αυτέ τι διαφορέ, εργονομική ε, κίνδυνη παραδοσιακή παραδοσιακή που πρέπει να αντιμετωπίζουν στην εργασία του οι εργαζόμενοι. Μπορούμε να δούμε από το ερωτηματολόγιο ότι όσο περισσότερο εκτίθενται σε οικονομικού, σε, με συγχωρείτε, σε κινδύνου όσον αφορά για παράδειγμα την το να σηκώνουν μεγάλα βάρη ή να έχουν ε, ε, προβλήματα όσον αφορά την, ε, τον κλονισμό που τους προκαλείται σωματικά, όλο και λιγότερο θα θεωρούν ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Επίσης, όσον αφορά την διασφάλισή τους σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εκείνοι που έχουν την μεγαλύτερη ένταση, το μεγαλύτε τη μεγαλύτερη πίεση σε σχέση και με την αυτονομία τους, πολύ λιγότερο θα μπορούν να απαντήσουν καταφατικά ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με τα καθήκοντά τους στα 60 τους χρόνια. Αν συγκριθούν με εκείνους που απασχολούνται σε λιγότερο απαιτητικέ θέσεις απασχόλησης ή εκείνους που έχουν μεγαλύτερη αυτονομία κατά την εργασία τους. Και πάλι αυτό το οποίο πιστεύουν οι εργαζόμενοι ότι θα είναι σε θέση να κάνουν ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στα ποσοστά που πραγματικά βρίσκουμε ηλικιακά ε, ε, στο εργατικό δυναμικό. Πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπίσει. Φυσικά το να αλλάξει η διοργάνωση της εργασίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να δεχτούμε. Όμως εγγενώς υπάρχουν κάποιες ε, επιπτώσεις της ε, μεγαλύτερης έντασης. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχει άλλη αναλλακτική λύση για ένα εργαζόμενο από το να αλλάξει ε, απασχόληση, θέση εργασίας ή να αποχωρήσει από το, την εργασία τους. Και αυτό σε σχέση με εκείνους που αντιμετωπίζουν μια τέτοια προοπτική είναι σαφές ότι έχοντας καταρτιστεί σε τακτά διαστήματα στη ζωή τους ε, κατά τη διάρκεια της αδειοδρομίας τους βοηθά να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε στο ερωτηματολόγιο αυτό ότι η πρόσβαση στην κατάρτιση με την ε, αυξανόμενη ηλικία ε, ακολουθεί ένα αυθύνοντα ρυθμό και μεταξύ των 30 και 49 μικρότερο ποσοστό εργαζομένων που έχουν ε, ε, λάβει κατάρτιση. Αυτό μειώνεται σε 30% για εκείνους που είναι πάνω από 50 ε, ετών στην ηλικία τους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως από την άλλη πλευρά ότι πολλά έχουν γίνει για να βελτιωθεί η ποιότητα στους χώρους απασχόλησης και από τις επιχειρήσεις. Και γνωρίζουμε ότι προβληματίζονται και επενδύουν οι εταιρείε όσον αφορά στην, την ποιότητα στην εργασία όχι για κάποιους ε, λόγους ε, ε, φιλανθρωπίας, αλλά επειδή αναμένουν να υπάρχουν κέρδη και ωφέλη για την εταιρεία τους. Πρόσφατα είχαμε μια μελέτη περιπτώσεων σε εταιρείε για να δούμε αν και κατά πόσον αυτή η διασύνδεση μεταξύ ποιότητα στην εργασία και επιδόσεων υφίσταται και τα αποτελέσματα είναι αρκετά σαφή. Είναι σαφές πλέον ότι η διασύνδεση, η σχέση μεταξύ κατάρτισης δεξιοτήτων, απασχολησιμότητας και επιδόσεων είναι ισχυρή. Η κατάρτιση βελτιώνει την επίδοση και δημιουργεί δυνατότητες να χρησιμοποιείται τεχνολογία αλλά και να αυξηθεί η ικανότητα να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Επίσης υπάρχει σαφής διασύνδεση σε σχέση με την προώθηση της σταδιοδρομίας και των δεξιοτήτων και όσον αφορά των πολιτικών για την αντιστάθμιση των ε, ε, διαφορετικών αυτών προσεγγίσεων. Θα μπορούσε κανείς να ακολουθήσει αυτή την πορεία και να πάει ένα βήμα παραπέρα και να πει αν εταιρείε χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους διαχείρισης όσον αφορά τον ελαστικό χρόνο απασχόλησης, ε, την δυνατότητα κατάρτισης, δεν θα έπρεπε να διασφαλίζουν ένα υψηλότερο ποσοστό ποιότητας αλλά και την βελτίωση των όρων απασχόλησης για τους εργαζομένους και πάλι το εξετάσαμε και καταδεικνύεται ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις ε, όταν αυτές οι πρακτικές ε, εφαρμόζονται σε εταιρείε που έχουν πάνω από τον μέσο όρο παραγωγικότητα, παραγωγικότητα κατά τα τελευταία χρόνια, τρία χρόνια και καλύτερη οικονομική κατάσταση και επιδόσεις. Μπορούμε να δούμε δηλαδή ότι η καλύτερη έκβαση για τους εργαζόμενους συνδέεται με την καλή διοργάνωση εργασιακά από πλευράς της εταιρεία και αυτό εκφράζεται και στατιστικά. Ευχαριστώ τελευταίος παρεμβαίνων είναι ένας ε, ε, ειδικό για τα θέματα της αγοράς εργασίας, ο καθηγητής Μάικλ Κάμπελ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι χαρά μου που βρίσκεται εδώ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω την τελευταία 20 ετία της ζωής μου σε έξι λεπτά. Ε, αυτή η ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας είναι ζωτική σημασίας, κρίσιμη σημασίας και χαιρετίζω ενθουσιοδός την έκθεση της Κομισιόν. Ελπίζω ότι αυτά που θα πω τα επόμενα λεπτά θα προσθέσουν κάποια αξία σε αυτή την ε, έκθεση. Θα επικεντρωθώ στη σχέση μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασία αλλά αυτά που θα πω έχουν σχέση και με την γενικότερη λειτουργία της ε, αγοράς εργασίας, την ευελιξία με ασφάλεια, τη χρήση του εργατικού δυναμικού που ανέφερε και η Μπάρμπαρα και την ε, αναβάθμιση της ποιότητας των θέσεων εργασίας. Ας πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Αν σκεφτείτε ότι έχει προβλήματα η Ευρώπη σήμερα, στο μέλλον θεωρώ ότι θα έχουμε μεγαλύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες όμως ταυτόχρονα, γιατί όλες οι προκλήσεις μπορούν να μεταφραστούν σε ευκαιρίες με τη σωστή δράση. Ουσιαστικά υπάρχουν μεγάλες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην οικονομία, την αγορά εργασίας, άρα και στις δεξιότητες που χρειάζονται με βάση τις δημογραφικές αλλαγές, τεχνολογία, τις κοινωνικές αλλαγές. Αυτό το διάγραμμα είναι μια μικρή σύνοψη όλων αυτών, μιας έκθεσης δηλαδή 200 σελίδων. Ουσιαστικά, οι περισσότερες αλλαγές ε, επηρεάζουν τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για συμμετοχή στην αγορά εργασίας και για την επιτυχία της αγοράς εργασίας και βεβαίως ε, αυτά επηρεάζουν και τα, τους εργαζομένους και τους εργοδότες. Αν τα κάνουμε όλα σωστά θα κερδίσουν όλοι. Είναι από τα λίγα πράγματα που θα αποφέρουν κέρδος και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες. Ενώ όλοι θα χάσουν αν δεν τα κάνουμε σωστά. Επόμενο, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι σωστή η στρατηγική, σωστό το πλαίσιο και κατά δεύτερο λόγο θα σας εξηγήσω το διάγραμμα που το φτιάξαμε στην οργάνωσή μου όπου είμαι 8 χρόνια είναι η Βρετανική Επιτροπή Απασχόλησης και Δεξιοτήτων. Σας τη συστήνω όχι γιατί είναι Βρετανική οργάνωση αλλά πραγματικά πιστεύω ότι έκανε πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά σε αυτό το τομέα. Η δουλειά μας είναι να συμβουλεύουμε τις κυβερνήσεις της ε, Βρετανίας σχετικά με πρόοδο στις δεξιότητες και θέσεις εργασίας και τι πρέπει να κάνουν εκείνοι μετά σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα επικεντρωνόμεθα στην ε, βελτίωση των επενδύσεων του εργοδότη που είναι κρίσιμο θέμα για την επιτυχία όπως θα δείτε. Εμείς είμαστε ανεξάρτητος φορέας, αυτό είναι σημαντικό. Οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στον φορέα μας και χρηματοδοτούμεθα από το δημόσιο ε, είμαστε ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση όμως και έτσι μπορούμε να κάνουμε ριζοσπαστικές προτάσεις αλλαγέ, για αλλαγές. Οι δεξιότητες είναι σημαντικές για την ανάκαμψη προφανώς, αλλά είναι μια άβολη αλήθεια το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχετικά χαμηλές δεξιότητες. 7 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ή έχουν χαμηλή εξειδίκευση και δεν μπορούν να εργαστούν στην αγορά εργασίας του 2020, το 1 τρίτο όλων των ενηλίκων δηλαδή. Χρειάζεται πλαίσιο λοιπόν. Πρώτα θα πρέπει να δούμε την έκβαση, την ε, ευημερία και ποιο είναι, ποια είναι η τελική έκβαση. Μεγαλύτερη ευημερία, παραγωγικότητα, δηλαδή ε, εισοδήματα, απασχόληση και μεγαλύτερη ισότητα. Και με τρεις τρόπους θα γίνει αυτό. Πρώτα θα αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες, καλύτερη προσφορά καλών δεξιοτήτων και καλύτερη σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων που έχουμε και των δεξιοτήτων που χρειαζόμαστε. Δεν έχει νόημα από οικονομικής άποψης να ε, προσφέρουμε δεξιότητες που δεν έχουν ζήτηση. Είναι μεγάλη απογοήτευση αυτή και δημιουργεί και αγανάκτηση στον κόσμο. Τρίτον και τελευταίο, και συχνά αυτό λείπει στο παζλ μας, θέλουμε να έχουν περισσότερες ε, φιλοδοξίες οι εργοδότες, γιατί σε τελευταία ανάλυση οι θέσει εργασία και δεξιότητε εξαρτώνται από τη συμπεριφορά των εργοδοτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ατζέντα των θέσεων εργασία. Οικονομική πολιτική, πολιτική αγορά εργασία, πολιτική εκπαίδευση κατάρτιση. Αυτά θα συνδεθούν για να προχωρήσουμε. Και κάτω στο διάγραμμα, για να το θυμόμαστε όλοι, μιλάω για το πούμα που είναι ένα πολύ χαριτωμένο και όμορφο ζώο, αλλά αυτό εδώ είναι ένα ε, ε, ε, ακρονίμιο, δηλαδή ευημερία, αναβάθμιση, αντιστοιχία και φιλοδοξία στα αγγλικά. Προχωρούμε λοιπόν. Στα γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Εδώ ένα διευρυμένο διάγραμμα αυτού που είδατε, το προσπερνώ, πάμε στο επόμενο. Θέλω να πιάσω κάθε συνιστόσα που συμβάλλει στην ευημερία, δηλαδή η αναβάθμιση, η αντιστήχηση, η φιλοδοξία. Ένα λεπτό θα αφιερώσω στην καθεμία για να δείξω ποιο είναι το βασικό εργαλείο επίλυσης του προβλήματος. Καταρχήν θα πρέπει να δείξουμε τα πλεονεκτήματα για την εκπαίδευση, ε, κατάρτιση, εξειδίκευση. Να ενθαρρύνουμε Περισσότερου ανθρώπου, εταιρείε να επενδύσουν σε δεξιότητε, Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίε, θα τα πούμε σε ένα λεπτό αυτά. Μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά εργασία και καλύτερο προσανατολισμό τον νέων επαγγελματικό προσανατολισμό. Το σύστημα εκπαίδευση κατάρτιση από τα ε, σχολεία, πανεπιστήμια, κολέγια να είναι υψηλή ποιότητα και να βεβαιωθούμε ότι αυτά που κάνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έχουν σχέση με τη μετέπειτα ζωή των ανθρώπων και τι εμπειρίε του. και υπό αυτή την έννοια είναι σημαντικό να συμμετέχουν και οι εργοδότε. Και μετά να επεξεργαστούμε ποια είναι τα εργαλεία πολιτικής που είναι πιο πιθανό να βοηθήσουν στις αυξημένες επενδύσεις των εργοδοτών. Δεν μπορώ να τα συνοψίσω όλα βέβαια, αλλά δεν χρειάζονται όλες οι επενδύσεις δημόσιε δημόσιες χρηματοδοτήσεις μεγάλες. Και σε εποχή λιτότητας πρέπει να εντοπίζουμε τα μέτρα που είναι καλά από άποψη κόστους ωφέλειας. Και τα δίκτυα των εργοδοτών είναι ένα καλό εργαλείο γιατί είναι φθηνά οικονομικά και αποτελεσματικά. Ε, ένα, μια άλλη δέσμη θεμάτων είναι η αντιστοίχηση, δηλαδή δεξιότητες σε σχέση με ε, αυτά που χρειάζονται να κλείσουμε τα κενά σε δεξιότητες και να μειώσουμε την υποαπασχόληση και τη διαρθρωτική ανεργία που είναι πολύ υψηλές και ιδίως στην Ευρώπη. Να επικεντρωθούμε δηλαδή στις οικονομικά πολύτιμες δεξιότητες όπως τις λέμε και όπως είπα πριν οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας ε, παντού, όπως κάνει το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, δημιουργεί ε, τη δυνατότητα να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε σωστά τις πληροφορίες που έχουμε. Δεν είναι μόνο θέμα διαθέσιμης πληροφορίας, αλλά και αξιοποίησης της. Ε, θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν κατανοητά και να αξιοποιηθούν. Τώρα, ε, θα έλεγα να επικεντρωθούμε περισσότερο στην έκβαση, στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό ε, είναι σημαντικό, θα πρέπει να δώσουμε όθηση στην ατζέντα αυτή με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ας πούμε ε, πώς ανταμείβονται οι παρέχοντες εκπαίδευση από την επιτυχία των φοιτητών σπουδαστών που θα μπουν στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν πειράματα στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα σε σχέση με το ζήτημα αυτό και βέβαια οι διαμεσολαβητές, δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, ε, τομεακά συμβούλια είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, περισσότερες φιλοδοξίες. Ε, είπα ότι η ζήτηση για θέσεις εργασίας είναι μια παράγωγη ζήτηση, όπως λέμε, δεν παίζει μόνο ρόλο το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και η οικοδομική δομή θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες ισορροπίες. Είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε σωστά. Ε, ε, θα πρέπει, όπως είπε η Μπάρμπαρα, να δούμε το εσωτερικό της επιχείρησης. Χρειάζεται ε, καλύτερη, καλύτερο management, ε, ηγετικές ικανότητες, υψηλή απόδοση, αξιοποίηση των δεξιοτήτων που υπάρχουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος, αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά μαζί στην επόμενη διαφάνεια, ξαναγυρίζουμε στο πούμα. Ποια είναι η απόλυτη προτεραιότητα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες. Χρειάζεται να συμφωνήσουμε στην ατζέντα, θα πρέπει να ε, έχουμε ισχυρή δέσμευση, η κοινωνικοί εταίροι, οι κυβερνήσει των κρατών μελών, η Κομισιόν βέβαια και όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς. Χρειάζεται συνεχιζόμενη δέσμευση, ε, χρειάζεται μια νέα κοινή λογική για την ηλική μας. Όπως είπε και ο Βολτέρος, η κοινή λογική δεν είναι τόσο κοινή σε τελευταία ανάλυση και εγώ το έχω δει αυτό εκ πείρας. Νέα κοινή λογική της εποχής μας, αν την ε, εντοπίσουμε και αυτό είναι παράγον επιτυχίας, να συνδέσουμε τον κόσμο της ε, εκπαίδευσης, της απασχόλησης, ε, της οικονομίας, να δημιουργήσουμε ένα κύκλο αρετής, όπως είπα, μεταξύ της προσφοράς, της αντιστοίχης, της φιλοδοξίας, ε, θα πρέπει να ε, δούμε ε, πώς θα παρακολουθούμε την πρόοδο στα πλαίσια της στρατηγικής 2020, να είναι υπόλογα τα κράτη-μέλη, να κάνουμε κάθε φορά εκθέσεις πρόοδου. Δεν μπορούμε να πετάμε τα χρήματα, του, τα κρατικά κονδύλια. Σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη αλλαγή, συνεχιζόμενη αλλαγή στην ε, νοοτροπία και τη συμπεριφορά εργοδοτών και εργαζομένων. Υπάρχουν πολλοί οικονομικοί τρόποι για να γίνει αυτό με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Δεν χρειάζονται δηλαδή τεράστια κονδύλια. Και τέλος, αυτό το η διαφάνεια μας θυμίζει γιατί κάνουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί ένα εργατικό δυναμικό με πτωχές δεξιότητες δεν κάνει φτωχότερη τη ζωή των εργαζομένων, αλλά τη ζωή όλων μας. Έτσι λοιπόν η ψηλή εξειδίκευση σε εργατικό δυναμικό δεν εμπλουτίζει μόνο τις δικές τους ζωές αλλά τις ζωές όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση που μας έκανε πλουσιότερους. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια στο τέλος, η κυρία Γιαζοβίτσκα και μετά η κυρία Μογά. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε σχέση με την παρέμβαση για την αγορά εργασίας και το θέμα της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά εργασίας είναι σημαντικό και η στρατηγική που ανέφερε ο καθηγητής Κάμπελ. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να αλλάξουν τα πράγματα. Θα ήθελα μια πληροφορία που είδατε απουσιάζει και που σχετίζεται με τα βέλτιστα καλά παραδείγματα, πρότυπα, για παράδειγμα, για διάφορα ιδρύματα, για το ε, ίδρυμα ε, που ασχολείται με θέματα μελετών ε, εργαζομένων και εργοδοτών. Δεν υπάρχει κάποια ξεχωριστή σύσταση. Αν δεν υπάρξει συνεργασία όμως μεταξύ των διαφορετικών ιδρυμάτων και φορέων, θα καταλήξουμε στο να μην υπάρχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Η κυρία Μωρέν και μετά ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς και την κυρία Μπάστος που οργανώσατε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Έχουμε ένα ουσιαστικό πρόβλημα και θα ήθελα να επισημάνω δύο ή τρία σημεία τα οποία είναι πολύ προβληματικά. Το πρώτο θέμα είναι η άνοδος, η ανοδος άνοδος των προδιαγραφών. Και αυτό βέβαια έχει αμέσως σχέση και με τις μελλοντικέ θέσεις εργασίας, γιατί θα αλλάξουν και οι θέσεις εργασίας και πώς είναι δυνατόν εμείς ε, να ε, αυξήσουμε και το επίπεδο των προδιαγραφών και από την άλλη να αντιμετωπίσουμε την εξέλιξη των θέσεων ε, εργασίας ανά επαγγελματικό κλάδο. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που θα τεθεί σε όλες τις ε, χώρες και πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε. Το δεύτερο ζήτημα είναι πώς θα κινητοποιηθούμε παρά το ε, ε, δεδομένου ότι ο χρόνος ε, εργασίας και ο χρόνος των προδιαγραφών δεν είναι ίδιος. Ο χρόνος της εκπαίδευσης, της κατάρτισης είναι πάντα μεγαλύτερος και πώς είναι δυνατόν συνεπώς να είναι πιο αποτελεσματική η δράση. Τρίτον, ε, άκουσα την, ε, την άποψη για, τα, για τους ε, εκπαιδευτές. Το βασικό που πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτής είναι να μπορεί να εκπαιδεύει τους πάντες. Γιατί Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ε, για εκπαιδευτές οι οποίοι ε, θα ασχοληθούν κυρίως ε, με τους ανθρώπους με περισσότερες προδιαγραφές και κανένας δεν θα θέλει να επικεντρωθεί σε αυτούς που, έχουν τις μεγαλύτερη, που έχει τη μεγαλύτερη δυσκολία εκμάθησης που είναι οι άνθρωποι χαμηλότερης, χαμηλότερων προδιαγραφών. Ο κύριε Κρίστανσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι ε, μπορεί κανείς να μακρηγορήσει. Μια πολύ σύντομη ερώτηση έχω. Κάνετε λόγο για την flexicurity. Συχνά, αν δει κανείς όμως τι συνέβη με την flexicurity τα τελευταία χρόνια, μπορεί κανείς να δει μια πολύ μεγάλη αύξηση στις επενδύσεις στην ελαστικότητα και μείωση στην ασφάλεια. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε την ορθή ισορροπία μεταξύ των δύο στοιχείων της Flex Security. Είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στον τομέα της ασφάλειας. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει απλά η ευελιξία. Το βλέπουμε και από τη χώρα μας ε, στην Δανία αν υπάρχει η προοπτική του να γίνει κάποιος ε, άνεργος, υπάρχουν επιδόματα ανεργίας, μπορεί κανείς ε, να μετακινηθεί και να δει στην αγορά εργασίας ποιε δυνατότητες υπάρχουν μέσω της δυνατότητας για την ασφάλεια αυτής της συνιστώσας. Μπορείτε να τοποθετηθείτε επ' αυτού. Η κυρία Μπάστος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις που έγιναν από τους ε, ε, πραγματογνώμονες και πρέπει να πω ότι έχω και ένα μέλημα, μια ανησυχία σε σχέση με την πλαισίωση της κρίσης ε, που, στην οποία βρισκόμαστε και αυτή την αφετηρία ως σημείο που έχει επιπτώσει σε όλα τα μέτρα και σε όλες τις ε, ε προτάσεις που γίνονται και που προβλέπονται σε σχέση με την εργασιακή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είμαστε παραγωγικοί, να είμαστε στο ύψος ε, των απαντήσεων που πρέπει να δοθούν στις προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και ε, κάτι το οποίο ε, ε, τονίστηκε για τις κοινωνικές πολιτικές για την απασχόληση που πρέπει να ακολουθηθούν τα επόμενα χρόνια για να προσαρμοστεί η αγορά εργασίας σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν και τις ελλείψεις που είναι πολύ σημαντικές Επίσης να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευθεία στην ε, προσέγγιση και μεγαλύτερες επενδύσεις ε, όσον αφορά την κατάρτιση και τα αναγκαία μέτρα που είναι αναγκαία για να βοηθηθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη. Ο κοινωνικός διάλογος επίσης και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να αναζητηθούν στις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Επίσης σημειώνω ότι εκκινώντας από ένα σημείο το οποίο είναι συνενετικό θα έλεγα μεταξύ μας σε σχέση με τις συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας και περικοπών στα κράτη-μέλη, δεν πρέπει να χάσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας, το φιλόδοξο πλαίσιο για να δράσουμε, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης με καλύτερη ποιότητα, με μεγαλύτερα προσόντα για να πετύχουμε να ανταποκριθούμε στο ε, ενδυνάμει δυναμικό αύξησης ε, και το, το ανθρώπινο δυναμικό και τις ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι ευχαριστώ όλους τους πραγματογνώμονες. Μήπω θέλει κανεί από του προσκεκλημένου να απαντήσει στο ερώτημα του κυρίου Κρίστενσεν. Κύριε Κάμπελ, όχι. Η κυρία Γερστενμπέργκερ. Θα προσπαθήσω, δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα τα καταφέρω. Ένα που θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με τη συζήτηση για τα θέματα flexicurity και την flexicurity στα θέμα, στην περίοδο κρίσης είναι το παράδειγμα της μερικής απασχόλησης, γιατί εκεί υπάρχει ο συνδυασμός ε, ε, ελαστικότητας αριθμητικής για τις ανάγκες μιας επιχείρησης και ταυτόχρονα απασχόληση και διασφάλιση εισοδήματος για τους εργαζόμενους μικρότερη απασχόληση, καμιά φορά και σε μηδενικό χρόνο απασχόλησης, όμως από την κατάσταση αυτή διασφάλιση σε σχέση με το επίπεδο ε, ε, ε, των εργασιακών απολαβών. Εκείνο το οποίο βλέπουμε να απουσιάζει από αυτά τα, από αυτά τα σχέδια είναι το στοιχείο της κατάρτισης που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση δεξιοτήτων. Φυσικά τέτοιου είδους μαθήματα κατάρτισης και επιμόρφωσης πρέπει να προσαρμόζουν και να δίνονται κάτι ομαδοποιημένα, γιατί κανείς ποτέ δεν μπορεί να ξέρει επί πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα διατηρηθεί η περίοδος μερικής ή μικρής ε, περιορισμένης απασχόλησης, αλλά επίσης και στην πλευρά των επιχειρήσεων να ταυτοποιηθούν εκείνοι οι οποίοι θα είναι ε, δυνατόν να καταρτιστούν. Το είδαμε αυτό στην έρευνά μας. Ένα ευάλωτο στοιχείο από τα θετικά ε, τα οποία έχουμε ως αποτελέσματα για την flexicurity στην περιορισμένη απασχόληση είναι η περιορισμένη δυνατότητα χρήσεως τέτοιων ευκαιριών για την κατάρτιση. Ευχαριστώ. κύριος Βισεντίνη παρακαλώ. Για αυτή την τελευταία παρέμβαση ε, της, της, της ειδικού, ακριβώς το ίδιο ήθελα να πω κι εγώ. Πολύ λίγες χώρες έχουν εφαρμόσει την ε, Flexi Security συνδυάζοντας την, ε, πραγματικά την ευελιξία και την ασφάλεια. Διότι πριν από την κρίση στην μεγάλη πλειοψηφία των ε, χωρών υπήρχαν οι ευάλωτες αν θέλετε, θέσεις εργασίας και μετά την κρίση η κατάσταση επιδεινώθηκε χωρίς να υπάρχει ε, προστασία των ε, εργατικών δικαιωμάτων και των θέσεων απασχόλησης που συνεχίζαμε να, χάσουμε, να χάνουμε και προφανώς δεν βοήθησε κανείς τους εργαζομένους ε, σε αυτές τις θέσεις απασχόλησης που δεν ήταν καθόλου σίγουρες και ασφαλείς θα πρέπει να συνδυάσουμε την παρέμβαση των επιδοτήσεων που είναι σε μια περίοδο κρίσης θα πρέπει να αυξάνονται και όχι να μειώνονται. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η πολιτική των περικοπών των κοινωνικών ε, δικαιωμάτων πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, θα πρέπει να αυξήσουμε τις επιδοτήσεις, αλλά ταυτόχρονα μαζί με, τα, με τις επιδοτήσεις ή τα επιδόματα θα πρέπει να ε, ε, βοηθήσουμε για να καταρ... Ε, έτσι ώστε να καταρτίζονται καλύτερα οι εργαζόμενοι. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων που η θέση τους είναι επισφαλής στην αγορά εργασίας. Για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό και να, συντο... να, να συνδυάσουμε αν θέλετε τις ανάγκες ε, ε, και των ε, επιχειρήσεων για κατάρτιση θα πρέπει να υπάρξει ένας κοινωνικός διάλογος, ένας ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος ανάμεσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών. Διότι μόνο ανάμεσα σε ένα, μέσα από έναν διάλογο μπορούμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες κατάρτισης που απαιτεί η αγορά εργασίας, να ε, καλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν και να, μέσα από τις κοινέ ανάγκες των εργαζομένων και των εργοδοτών να προσφέρουμε στις δημόσιες αρχές σε κρατικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την, ε, την κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των εργαζομένων. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση έκανε πιο δύσκολες τις σχέσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και ε, έχει αποδυναμώσει τελείως τον κοινωνικό διάλογο, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε επίπεδο κρατών. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι απαραίτητος. Πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου για να επιληθούν όλε αυτές οι δυσκολίες. Επίσης, η κατάσταση έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, αυτό το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε τα προβλήματα κατάρτισης, ε, επαγγελματική κατάρτισης, ούτε τα προβλήματα της αγοράς, ε, αγνοώντας ε, την κατάσταση και να θεωρούμε ότι είμαστε όπως ήμασταν πριν από την κρίση. Αυτές, ούτως ή άλλως αυτές οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν είχαν ξεκινήσει πριν από την οικονομική κρίση. Άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα εργαλεία μας σε αυτή τη τελείως νέα αγορά εργασίας. Διότι ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες κατάρτισης των επιχειρήσεων. Μάλιστα, ωραία. Ολοκληρώσαμε με την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Ε, θα ήθελα ε, να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλό κουράγιο στην εισηγητριά μας. Στις 12 και 13 Ιουλίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες της και ελπίζω ότι θα μας έχει τροφοδοτήσει η σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους μας. Η Business Europe δεν θέλησε να συμμετέχει στην συζήτησή μας. Ευχαριστεί η Πρόεδρος και τους διερμηνείς ε, που μας ε, που επειδή μας ε, οδήγησαν στο τέλος των εργασιών μας.